Αρχίζουμε με την ε, έγκριση της μερίσιας διάταξης. Θα ήθελα να σας πω, να σας μιλήσω για μία αλλαγή το σημείο 15. Α, έκανα λάθος. Καλή μας αρχή. πάντα μου κάνετε πλάκες. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, λέει η πρόεδρος. Okay. Donc Διαρθρωμένος διάλογος σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012. Η παρουσίαση των προτεραιοτήτων για, τις, ε, για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική το 2012 θα γίνει από τον Επίτροπο Άνδρης Πίμπαλξ. Μια μισή ώρα θα, για μια μισή ώρα θα γίνει η συζήτηση. Έτσι προβλέπεται διαρθρωμένος διάλογος λοιπόν για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2012. Θα θυμόσαστε ότι η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπή στον Οκτώβριο του 2010 επιτρέπει στους βουλευτές να προωθήσουν τις ιδέες τους για το επόμενο έτος. Επειδή η Επιτροπή δεν έχει ορίσει το πρόγραμμα εργασίας για το 2012 ή τουλάχιστον όχι ακόμα, θα ήταν σκόπιμο να συζητήσουμε τώρα την αναπτυξιακή πολιτική και τους τομείς που θα πρέπει να μας απασχολήσουν του χρόνου θα συζητήσουμε όλες τις πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου για το επόμενο έτος και μέχρι το τέλος, μάλλον πριν από το τέλος του έτους, θα λάβουμε την πρόταση κανονισμού που θα αντικαταστήσει το μέσο για την αναπτυξιακή πολιτική που λύγει το 2013. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε όλα τα θέματα και ως προς τα έγγραφα μη νομοθετικού περιεχομένου όπως την Πράσινη Βίβλο και τις ανακοινώσεις και μετά τη λήξη τη συνεδρίασης οι συντονιστέ θα φτάσουν σε συμπεράσματα μαζί με τον Επίτροπο και θα προβούν προς που θα αποστείλουν προ τη διάσκεψη προέδρων των Επιτροπών για τι προτεραιότητε για το 2012. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Πίμπαλξ. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη η δονή που αισθάνομαι σήμερα για αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τον δομημένο που λέμε διάλογο. Η αναπτυξιακή μας πολιτική έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων θα πρόκειται για ένα πολιετές πλαίσιο και σήμερα θα μιλήσουμε για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Πιστεύω ότι η αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Είμαστε αποφασισμένοι να εξυγχρονίσουμε την έννοια αυτή της ανάπτυξης, να είναι πιο στοχευμένη, πιο αποτελεσματική και πιο αποφασιστική. Και θέλω η Κομισιόν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της. Δεν είναι κάτι το εύκολο, γιατί απαιτούνται αλλαγές πολλών στοιχείων και οι αξιολογήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου που συνήθως έχουν είναι θετικές κάνουν μερικές φορές ορισμένες χρήσιμες συστάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων προγραμμάτων. Μερικές φορές η απάντησή μας πρέπει να δοθεί, να βρεθεί μέσα σε μια πολύ πολύπλοκη πολιτική ατμόσφαιρα. Παραδείγματος χάρη είχα συναντήσει πριν έρθω εδώ εκπροσώπους του Σουδάν. Τον Ιούλιο θα εγκαινιαστεί το νέο κράτος στο νότο του Σουδάν, αλλά υπάρχει πρόβλημα και ανατολικά του Σουδάν, στο Δαρφούρ. Πολλά προβλήματα λοιπόν και ε, δύσκολη πολιτική κατάσταση. Θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν πολλές προκλήσεις. Πιστεύω όμως ότι τελικά θα βασιστούμε στις διαδικασίες που προέβλεπε η πράσινη βίβλος που έφερε τον τίτλο «Πώς να προχωρήσει η αναπτυξιακή μας πολιτική». Όλοι νομίζω λίγο πολύ μπορούμε και πρέπει να συνυπογράψουμε τέτοιες προτάσεις γιατί ο στόχος μας θα είναι κυρίως η μεγαλύτερη αποτελεσματικότης και όχι μόνο στα χαρτιά. Έτσι θα διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε δαπανάτε για να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες θα προβλέπονται και έγγραφα μεμονωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών αναχώρα. Τέλος, θα εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για στήριξη από τον προϋπολογισμό ή του προϋπολογισμού που αποδείχτηκε τελικά κάτι πολύ δημοφιλές. Θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε και με τις αξίες που συμμεριζόμαστε όλοι. Τις προτάσεις για την, το λεγόμενο budget support θα τις υποβάλουμε τον Σεπτέμβριο. Μετά θα συζητήσουμε το πιο δύσκολο θέμα από όλα, δηλαδή την πρακτική τους εφαρμογή. Και πιστεύω ότι έχουμε πολλά, χρειάζονται πολλά που πρέπει να γίνουν. Παραδείγματο χάρη για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν γύρω σε, πάνω σε μια κοινή άποψη σε συνδυασμό με τα μεμονωμένα αναπτυξιακά έγγραφα αναχώρα ε, δεν θα είναι κάτι εύκολο. Επίσης πρέπει να μιλήσουμε για τα θέματα του χρηματοδοτικού πλαισίου, που, του δημοσιονομικού πλαισίου που θα λειτουργεί μέχρι και το 12. Η καιροί είναι δύσκολη, αυτό το ξέρουμε όλοι και όλες καλά. Αλλά δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τις προσδοκίες μας. Υπήρξε η υπόσχεση του 0,7% του ΑΕΠ και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν για να πείσουμε τις χώρες μέλη για την ανάγκη να διατηρηθεί η στήριξή τους για την ανάπτυξη είμαι αποφασισμένος να αποδείξω, να τους δείξω ότι όλα αυτά μπορούν να αποφέρουν, να φέρουν αποτελέσματα. Τέσσερα στοιχεία θα μπορούσα να προτείνω. Πρώτον, να αναρωτηθούμε τι μπορεί να βελτιωθεί σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο η Κομισιόν θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ παραπάνω από τον 28ο Ευρωπαίο Δωρητή, να γίνει δηλαδή ο καταλήτης μιας γενικότερης συστημικής αλλαγής. Θα ήθελα να μην ξεχνάτε ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ένωσης είναι η δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες ε, και πιο ενιαίες εσωτερικές αγορές του κόσμου. Πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε την επιτυχία αυτή να την επιδείξουμε ως υπόδειγμα και στον αναπτυσσόμενο κόσμο ο οποίος ιδιαίτερα δε η Αφρική δεν εκμεταλλεύεται όλες του τις δυνατότητες στο έπακρο. Για ό,τι βοήθεια χορηγεί λοιπόν η Κομισιόν θα χορηγεί και μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας για καλύτερη οικονομική, για καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα και θα ζητήσω περισσότερο συνδυασμό των προγραμμάτων για την ανάπτυξη παραδείγματος χάρη για θέματα κατά πολέμης αντιμετώπισης των κλιματολογικών αλλαγών. Δεύτερον, πρέπει να χορηγηθούν μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα μέσω της χρήσης καινοτόμων νέων μεθόδων Ο προσόφελος φυσικά των πολιτών. Τρίτον, πρέπει όλες οι χώρες με αυστηρότερους προϋπολογισμούς να αποδείξουν ότι κάνουν παραπάνω από οποιονδήποτε άλλον δωρητή, ότι προσφέρουν παραπάνω από οποιονδήποτε άλλον δωρητή θα μπορούσαν όλα αυτά να αποτελέσουν έναν κινητήρα, κινητήρια δύναμη για την αλλαγή που θα βοηθούσε και την κάθε κυβέρνηση να βελτιώσει τις προσπάθειές της για δημοκρατική ανάπτυξη. Πρέπει όμως όλα τα υπάρχοντα εργαλεία να χρησιμοποιούνται με πιο στοχευμένο και επιλεκτικό τρόπο, παραδείγματος χάρη Έχω πιστεί ότι η στήριξη των προϋπολογισμών θα ωφελήσει μόνο τις χώρες που συμμερίζονται τις δημοκρατικές και βασικές μας αρχές. Και εκεί θα, μπορούσαν, θα μπορούσε αυτή η στήριξη όχι μόνο νομισματικά αλλά και με τις αξίες αυτές να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Πρέπει να δεχτούμε την απλή αυτή αλήθεια. Καμία αναπτυξιακή πολιτική δεν πρόκειται να πετύχει όπου δεν υπάρχει δημοκρατία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέταρτο, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες χώρες και να μεγιστοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνει η νέα συνθήκη της Λισαβόνας ώστε να παίξουμε πλήρως το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε διεθνώς και να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις διεθνώς. Γεωγραφικά σκοπεύω να κάνω μία ανάλυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων αναπεριφέρεια. Έχω σκοπό την εμπειρία που αποκτήσαμε από την περιφέρεια του Ειρηνικού να τη χρησιμοποιήσω και για την Κεντρική Ασία. θα δημιουργήσω έναν κατάλογο προτεραιοτήτων ως προς τις περιφέρειες και θα ζητήσω βελτίωση της υπολογισμότητας γιατί για να επιτευχθεί ο στόχος του 0,7% μέχρι το 2015 πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος. Ο ΣΑ πρόσφατα δημοσίευσε τα στατιστικά του στοιχεία και από εκεί φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντική η κατάσταση, είναι ενθαρρυντικά τα πράγματα. Δείχνουν τα στοιχεία αυτά ότι σε επίσημη βοήθεια έχουμε δαπανίσει 53,8 δισεκατομμύρια άρα πρόκειται για καθαρή επιτυχία το 10 αυτά αλλά δεν πετύχαμε την δαπάνηση του 0,56% του ΑΕΠ. Πολλές χώρες έχουν κάνει προσπάθειες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, ακόμη και η Πορτογαλία σημειώνουμε, τα σημειώνουμε λοιπόν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς άλλες χώρες βρίσκονται σε μεγαλύτερη καθυστέρηση και πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει συνέπεια. Και θα ήθελα να με βοηθήσετε εδώ για το θέμα των νέων χωρών μελών τις χώρες που μπήκαν μετά το 2004, από τις χώρες που μπήκαν μετά το 2004 μόνο η Κύπρος έχει πετύχει αυτό το στόχο του 0,56%. Όλες οι άλλες βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο και θα ήταν παρεξήγηση να θεωρήσουμε ότι ότι είναι αδύνατον να πετύχουν και οι υπόλοιπε χώρες τουλάχιστον αυτό το ποσοστό και να μένουν στο 0,23% κατά μέσο όρο που έχουμε διαπιστώσει. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική θέληση και ηγεσία γιατί αργότερα θα χρειαστεί να δαπανίσουν οι χώρες αυτές που βρίσκονται σε καθυστέρηση πολύ περισσότερα μετά για, για ανθρωπιστική βοήθεια ή στρατιωτικές παρεμβάσεις. Σχεδόν όλες λοιπόν οι νέες χώρες μέλη πρέπει να συνεχίσουν να τις σκληρές τους προσπάθειες και εγώ πρέπει να τους εξηγήσω καλύτερα γιατί όλα αυτά είναι απολύτως απαραίτητα. Σας είπα όμως ότι η κατάσταση δεν είναι απογοητευτική. Μπορώ λοιπόν να δώσω μια ενθάρρυνση σε, όλους, σε όλες τις χώρες Μερικές χώρες πρέπει να βελτιώσουν την κατάστασή τους, αλλά όλες μπορούν να το πετύχουν το στόχο. Κυρίες και κύριοι, το 2012 δεν θα χρειαστεί, δεν θα απαιτήσει καινούργιες ανακοινώσεις από την Επιτροπή, θα είναι έτος δράσης και αποτελεσμάτων ελπίζουμε και θα τονίζει ιδιαίτερα το πρόγραμμα πλαίσιο Κατά τη διαδικασία αυτή ξέρω ότι δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα και πρέπει όχι μόνο να είναι σωστά τα επίπεδα των δαπανών αλλά να γίνεται και σωστά, να γίνονται και σωστά οι δαπανήσεις. Ακόμη ισχύει ότι υπάρχουν πολύ καλά προγράμματα αλλά δεν είναι πολύ αποτελεσματικά. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τις στρατηγικές μας επιλογές. Πράγματι σήμερα η παρουσίασή μου δεν σας ανέφερε πολλές καινούργιες πρωτοβουλίες γιατί νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή της ήδη ισχύουσας διαδικασίας για εξυγχρονισμό και να πετύχουμε πραγματικές αλλαγές ιδίως με βάση την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την πολιτική εξυγχρονισμού. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τον εαυτό μας με όλο και καινούργια στρατηγικά προγράμματα, αλλά να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο τι έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται και να δούμε πώς θα μπορούσε αυτό να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους συντονιστές, αν το επιθυμούν. Ο κύριος Μίτσελ. Thank you, Madam President, and thank you, Commissioner. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση, κύριε Πίτρο. Πολλά κράτη-μέλη κάνουν, μάλλον παλινοδούν ως προς τον προϋπολογισμό και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Από όσο θυμάμαι, νομίζω ότι η Επιτροπή μίλησε για έξι δις ετησίως, δεν ξέρω αν ε, το αναφέρω σωστά, για να δούμε πώς θα πλαισιώσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό που έχει σημασία είναι να, είμαι πιο, να είμαστε πιο συντονισμένοι σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχει ε, ε, ε, μεγάλος αρνητισμός από τα κράτη-μέλη και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να το δούμε και μέσα στα πλαίσια της συνοχής. Ανθίστανται τα κράτη-μέλη λοιπόν, όπως είπα, και ίσως θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα και στη κοινή γνώμη των κρατών μελών. Εάν ο πληθυσμός δει ότι μπορούμε να έχουμε έξι δισετησίως με μεγαλύτερη συνοχή, θα το ήθελαν αυτό. Γιατί θα σώσουμε πολλές ζωές μικρών παιδιών, οι γυναίκες δεν θα πεθάνουν σε πολύ νεαρή ηλικία. Νομίζω ίσως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη γνώμη του κοινού. Σε σχέση με το έγγραφο για τις επιπτώσεις βλέπω ότι αναφέρονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση, η καινοτομία, τεχνολογίες, κλιματικές αλλαγές, ε, Yesterday, I'm very impressed Βιοπικιλότητα κλπ. Νομίζω ότι αυτό που διαπιστώνει τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα τα κινητά από ότι εγώ. Θα πρέπει λοιπόν να τα εξοπλίσουμε και για να τα εξοπλίσουμε θα πρέπει να διαθέσουμε κεφάλαιο. Θα ήθελα να θέσετε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Το συζητήσαμε αυτό στην Επιτροπή. αν έχουν, μάλλον αν ενισχύσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τότε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ε, ριζωθούν κάπου, να εγκατασταθούν κάπου. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πώς μπορούμε να το προωθήσουμε ε, αυτό. Πώς μπορούμε να δούμε και το ιδιοκτησιακό και να το προωθήσουμε. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό θέμα. Στην Αφρική και ειδικά Γκάνα, Μαδαγασκάρη και Νότια Αφρική υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο αρμόζει στην Αφρική ή την Αυστραλία και υπάρχουν ε, ε, δύο ε, κατευθύνσεις συμφερόντων. Θα ήθελα να σχολιάσετε γιατί ίσως θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αυτά τα επιστημονικά προγράμματα στην Νότια Αφρική. Δεν θα το γνωρίζατε βεβαίως, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, αλλά ίσως θα μπορούσε να σας απασχολήσει, διότι έτσι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια κρίσιμη μάζα στον τομέα της πραγματογνωμοσύνης και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να το σκεφτόμαστε, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με projects που αφορούν την Αφρική και την Αυστραλία ιδιαίτερα. Ίσως, ε, αν θέλετε, θα μπορέσω να σας αποστείλω συγκεκριμένα στοιχεία. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήρθα αργά, κύριε Επίτροπε, και γι' αυτό θα ήθελα το κείμενο της ομιλίας σας, γιατί κάποια πράγματα δεν τα άκουσα. Θα είμαστε ευγνώμονες αν μπορούσαμε να το έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για το 2012, το πρόγραμμα εργασίας για το 2012. Η ομάδα μας θεωρεί προτεραιότητα, πολύ σημαντικό για το 2012, η Κομισιόν να καταρτήσει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διαφάνεια στις εξορρυκτικές βιομηχανίες. Στη ΣΥΠΑ υπάρχει ο νόμος DOS-FRANK ή FRANK-DOT-FRANK ο νόμος Τότ Φρανκ, ευχαριστώ Τζούντιτ, που απαιτεί από τις εξορυκτικές βιομηχανίες να είναι ξεκάθαρες στα προγράμματα έργα τους. Όχι μόνο πώς λειτουργούν στις χώρες, αλλά επί τη βάση των έργων. Φαίνεται ότι στη ΣΕΛ δεν αρέσει αυτό και πιέζει για παρόμοια ευρωπαϊκή νομοθεσία με βάση τις εκθέσεις των χωρών. Καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε τη σαφήνεια που ακολούθησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και να ζητήσουμε διαφάνεια επί τη βάση των έργων. Οι εξορρυκτικέ βιομηχανίες πληρώνουν τους φόρους όπως πρέπει. Συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις της δεούσα επιμέλειας. Πώς αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα και άλλα πολλά ακόμα. Και επειδή αλλάζει γρήγορα ο κόσμος και επειδή, και επειδή αυξάνεται η ανάγκη για πρώτες ύλε, πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και να μην δεχόμαστε απλά η Ευρώπη να επιδιώκει τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντά της για να πάρει τους πόρους που χρειάζονται οι βιομηχανίες. Θα πρέπει να επιτρέπει με δίκαιο τρόπο να συμμετέχουν ισότιμα όλες οι χώρες. Να μην παρέχει μόνο, αλλά να ε, υπάρχουν και ωφέλη για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, ελπίζω ότι κάτι θα συμβεί εδώ γρήγορα και τι χρονικό ορίζοντα βλέπετε για το χρονοδιάγραμμα. Ίσως κι άλλοι θέλουν να το θίξουν αυτό. Η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πολιτικό ε, δυνητικό της βάρος αυτό θα γίνει αν μιλάμε με μια φωνή και μεγιστοποιείται το πολιτικό βάρος ε, όταν ε, δώσουμε βάρος σε πολιτικά θέματα, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου στις χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής. Γιατί αν πριν από μια δεκαετία μιλούσαμε την με μια φωνή, δεν θα είχαν υπάρξει αρνητικές εξελίξεις και θα ήταν καλύτερη η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τη στάση μας και να βοηθήσουμε για παράδειγμα τις εξελίξεις και τα νέα κινήματα στην Αίγυπτο, στην Τινησία, είδατε στην Αιθιοπία πόσο υποκριτικό είναι όταν δεν ε, τα σώμεθα υπέρ των δημοκρατικών αξιών και το ίδιο ισχύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ε, ίσα δικαιώματα. Η Κίνα, η Ρωσία δεν ενδιαφέρονται για την ισοτιμία στα δικαιώματα. Εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει τη διαφορά και εκεί βρίσκεται η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες στις χώρες του κόσμου. Στα... Όχι, θα προσθέσω κάτι ακόμα. Πριν σας ευχαριστήσω να προσθέσω κάτι για τη συνοχή την πολιτική συνοχή στην ανάπτυξη. Με ανησυχεί η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ινδία γιατί μπορεί να ε, δημιουργήσει πρόβλημα στην ανταλλαγή γενώσιμων φαρμάκων. Ποιος ασχολείται με το θέμα, λαμβάνεται υπόψη, το θέμα αυτό των γενώσιμων, που δεν είναι μόνο γενώσιμα, είναι και προϊόντα αλληλείας, συνοχή για την ανάπτυξη. Είναι απέτηση τη συνθήκη αυτό. Ποιο είναι υπεύθυνο εμείς, έχουμε τον Σκαρ Κέλλερ που είναι ο δικός μας εισηγητής για αυτό το θέμα, αλλά ο αρμόδιος στην Κομισιόν ποιο είναι. Εσείς ε, το κοιτάτε το θέμα, είναι δική σας ευθύνη ή πιανού. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που είναι παρόν γιατί είναι απόλυτα διαθέσιμος ε, σε σχέση με άλλους που συμμετέχουν στην, στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είναι μέλη της ΕΙΕΔ. Θα να πω ότι συμφωνώ με την δημοσιονομική του προσέγγιση. Στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. όταν ακούσουμε αυτά που λέγονται σε άλλες επιτροπές για την υποστήριξη του προϋπολογισμού βλέπουμε ότι λέγονται διαφορετικά πράγματα. Χθες ήμουνα στην ΑΦΕΤ για... και θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να καταβληθούν πολλές προσπάθειες αμοιβές κατανόησης πριν γίνει ε, λόγος για δημοσιονομική υποστήριξη. Δυστυχώς είδα ότι ε, απέχει πολύ από αυτά που λέμε εμείς και δεν είναι και η μόνη Επιτροπή. Θα πρέπει και οι άλλοι να, να μας συμπαρασταθούν. Ας κάνουμε λοιπόν μία προσπάθεια διαπαιδαγώγησης. Το είδαμε το θέμα με την ΑΦΕΤ και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Χωρίς να θέλω να κακολογήσω τους συναδέλφους, γιατί δεν βρίσκονται στην ίδια θέση με μας. Για το 2012 μιλήσατε για επικέντρωση των προσπαθειών στα αποτελέσματα και μιλήσατε για την ε, για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής μας. Θα ήθελα να σας κάνω δύο υποδείξεις επ' αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα καινοτομίας και από ε, πλευράς επινόησης καθαρά. Και αυτό το λέω για πολλούς λόγους. Εμείς ε, βασιζόμαστε σε μία σειρά ε, αξιών μέσα στα πλαίσια της λήψης αυτών των, αγαθών δεν θα πρέπει μέσα στα πλαίσια αυτά να μην είμαστε πιο φιλόδοξοι. Και αυτό αφορά και τις ε, ε, δύο διασκέψεις που θα γίνουν. Η δεύτερη θα γίνει στο, στην Κωνσταντινούπολη με βάση τις δηλώσεις του Παρισιού και της Άκρα θα πρέπει να μην διασυνδέουμε τη βοήθεια σε αυτή την πτυχή. Θα πρέπει και άλλες χώρες να συνεργαστούν με την Αφρική και να συμμετάσχει και η Αφρική σε αυτά τα πλαίσια ως προς την διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει αφορά τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Το θέμα αφορά το εξής. Θα καταπολεμήσουμε τη φτώχεια παντού ή στις πιο φτωχές χώρες που έτσι κι αλλιώς είναι επιλέξιμες για ε, δημόσια βοήθεια. Αυτό σημαίνει Κίνα, η Ινδία αλλά και Βραζιλία οι οποίες έχουν, είναι αναδυόμενες χώρες και έχουν ε, αρκετά υψηλά εισοδήματα. Έχουν ολοκληρώσει την ε, πορεία ανάδυσης. Εάν δεν πείσουμε αυτές τις χώρες να κάνουν μία επανακατανομή του πλούτου μέσα στην επικράτειά τους, δεν θα έχουμε καταπολεμήσει τη φτώχεια, γιατί διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα. Γίνεται μία διάσκεψη, θα γίνει μία διάσκεψη πριν από αυτή της Κωνσταντινούπολης και το θέμα είναι τι θα γίνει με τη συνένεση της Ουάσιντον. Έχει θαυτεί οριστικά και τότε τι νόημα έχει να αντικατασταθεί. Ένα άλλο θέμα που θίξατε και μπορείτε να βασιστείτε σε μας ένα άλλο θέμα αφορά ένα ενιαίο μπλοκ με 28 συμμετέχοντες. Οπωσδήποτε θα έχουμε ε, έναν προϋπολογισμό, όχι όμως υψηλότερο από τον τωρινό. Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε και τα εθνικά και τα κοινοτικά μέσα, θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες επί του θέματος. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την ε, μικροπρέπεια που υπάρχει από τη μία και την άλλη πλευρά. Φιλόδοξο είναι το σχέδιο, πράγματι, αλλά θα πρέπει η Ευρώπη ως πρώτος παγκόσμιος φορέας να δώσει κατευθυντήριες γραμμές, να ορίσει τις προτεραιότητες και οι άλλοι να μας ακολουθήσουν. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και έχουμε κάθε λόγο να είμαστε φιλόδοξοι. Ο κύριος Ντέβα από τους Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε Επίτροπε και μας μιλήσατε σαφή γλώσσα. Μιλήσατε για 52,8 δις ευρώ που δαπανίσατε σε διάφορα προγράμματα. Πριν από λίγους μήνες είχατε έρθει θυμάμαι και μας είπατε ότι θέλατε να, επιτύ... να εντείνετε τα προγράμματα εξηλεκτρισμού στην Αφρική. Πράγμα πολύ ωραίο. Γιατί αυτό συνδέεται με πολλούς άλλους τομείς. Επίσης για την περιουσία και την καταχώρηση των περιουσιών σε επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες που παράγουν, επισκευάζουν, κάνουν σέρβις, αλλά δεν αποτελούν κομμάτι της επίσημης οικονομίας, γιατί δεν έχουν εγγραφεί σωστά στα Μητρώα. Οπότε οι απασχολούμενοι είναι, λειτουργούν ανεπίσημα, δεν προπληρώνουν φόρους, δεν συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα στοιχεία, δεν, έχουν, δεν μπορούν να κάνουν αγορές ενώ δημιουργούν απασχόληση. Καλό θα ήταν λοιπόν να επισημοποιηθεί μέσα από εγγραφή σε Μητρώα όλων αυτών των ε, επιχειρήσεων ε, Το λόγο έχει η κυρία Γκρέσ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Ε, κύριε Πίμπαλκ, σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα για άλλη μία φορά ε, να αποζητήσω σαφείς απαντήσεις από εσά σε τρεις ε, τομείς. Το πρώτο μας μεγάλο μέλημα αφορά τη νομοθετική συνέχεια που θεωρούμε απαραίτητη σε σχέση με δύο εκθέσεις, την έκθεση υποδήματα για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και της ε, κυρία Ζολή για την φορολογική διακυβέρνηση στις υποανάπτυξη χώρες. Ποια συνέχεια θα δώσει σε αυτές τις εκθέσεις από νομοθετικής πλευράς και τι πρωτοβουλίες θα λάβετε ως προς τη φορολόγηση, τα έσοδα της οποίας θα μπορούσαν να δοθούν στην αναπτυξιακή πορεία αυτών των χωρών, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Το δεύτερο μας μέλημα αφορά την διατροφική αλυσίδα. Την παρχή τροφίμων, εδώ έχουμε κερδοσκοπία, διαφοροποίηση τιμών, αύξηση τιμών και αυτό αφορά και την ΚΑΠ και την κοινή ε, αλλιευτική πολιτική. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να αναστρέψει αυτή την τάση και να διασφαλίσει το δικαίωμα διατροφής, ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών πολιτικών. Τέλος, ένα τελευταίο σημείο αφορά την εξωτερική διάσταση της ε, κοινωνικής πολιτικής. Στην Επιτροπή αυτή έχουμε εγκρίνει μία γνωμοδότηση που ζητά από την Επιτροπή να εντάξει μία κοινωνική ε, ρήτρα μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ έτσι ώστε, ώστε μέσα στα πλαίσια των προτιμησιακών συμφωνιών, μάλλον οι προτιμησιακές συμφωνίες να μην παραμείνουν νεκρόγραμμα και να είναι δεσμευτικές. Ποια συνέχεια θα δώσετε και τι θα κάνετε έτσι ώστε να μην παραμείνουν αυτές οι συμφωνίες νεκρόγραμμα. Ευχαριστούμε. Οι άλλοι συντονιστές δεν είναι παρόντες. Δίνουμε το λόγο στα μέλη. Ο κύριος Κάσμαν. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Κάσμαν. Οι περισσότεροι θα με πλήρωναν να κλείνω το μικρόφωνο όταν μιλάω. Οπότε χαίρομαι που η πλειοψηφία προς το παρόν τουλάχιστον θέλει να το έχω ανοιχτό και να συνεχίσω. Επίτροπε, δεν θα σας αφήσουμε ε, τόσο εύκολα να γλιτώσετε εδώ. Είχατε εξαιρετικό πρόγραμμα το περασμένο χρόνο, το οποίο με μεγάλη πολιτική δέσμευση και αφοσίωση συνεχίσατε και προωθήσατε και με τους συναδέλφους σας και με το Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια λοιπόν αυτό που θέλουμε να πάρετε μαζί σας φεύγοντας από εδώ είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι δεσμεύσεις με πρόσθετα μέτρα που πρέπει να αναλυφθούν. Κάποια σύντομα σχόλια πριν επισέλθω στις λεπτομέρειες αυτών. Είπατε ότι πρέπει να είναι ε, υπόλογα τα κράτη-μέλη για το 0,7 του ΑΕΠ. Οπότε χρειάζεται τις έκθεση που θα εξετάζει αν τα κράτη-μέλη όντως ε, έκαναν αυτό που πρέπει για τη δέσμευση αυτή. Και αυτό είναι μέρος των πολιτικών πιέσεων που θέλετε να ασκούνται. Και αυτό γίνεται με τις κυβερνήσεις μας. Τώρα, για τον 28ο δωρητή που θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Είμαστε ο μεγαλύτερος ε, ε με ενιαίος δωρητής στον κόσμο. Είναι απαράδεκτο όταν πηγαίνουμε στα Ηνωμένα Έθνη, θα το ξέρετε εσείς, στην ε, σύνοδο για τις ε, στόχους της καθόμαστε εμείς ως παρατηρητής και όταν ε, γίνεται ψηφοφορία για το καθεστώς της Ένωσης, οι συνάδελφοι στην ΑΚΕ μας καταψηφίζουν. Οπότε υπάρχει εδώ μια ανισομερή εταιρική σχέση με κάποιες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμεθα. Όχι μόνο χώρες ΑΚΕ. Για του ΙΣΑΚΕ μιλήσατε για τις, τα θεμελιώδη, αρχές και αξίες. Ξέρουμε όταν κάναμε τις αναδιαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ότι οι ΑΚΕ δεν μας παίρνουν στα σοβαρά. Στη Κοινωνική Επιτροπή λίγες εβδομάδες πριν στην ΑΚΕ ετέθη ένα θέμα από το Προεδρείο των χωρών ΑΚΕ που συζητήσαν το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Φαινόμενο το λένε, φαινόμενο της ομοφιλοφιλίας. Πρώτη φορά με λένε φαινόμενο, το παίρνω σκοπλιμέντο. Το συζητήσουμε αυτό και να δούμε και το πολιτιστικό πλαίσιο. Πρέπει να πω ότι κάθε μέλος ΑΚΕ ε, που ήταν παρόν αρνήθηκε να συζητήσει. Δεν είπαν ότι πρέπει το θέμα αυτό να συζητηθεί. Πρέπει να δούμε το γερμανικό μοντέλο. Αυτή τη βδομάδα είπαν ότι θα αναστείλουν τη δημοσιονομική βοήθεια στο Μαλάουι. Όχι μόνο για αυτό που θα σας πω, αλλά και για αυτό, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας των γυναικών. Παρόμοιος νόμος για την ομοφιλοφιλία γενικότερα προγραμματίζεται να περάσει ε, και αλλού. Αν δεν ε, υπερασπιστούμε τις αξίες που προεσβεύουμε, πάντα θα είναι άνηση η σχέση και θα ακολουθήσουμε το δρόμο των Κινέζων ε, που περιορίζονται μόνο στην ανταλλαγή προϊόντων. Και περνώ έτσι στο θέμα που έθεσε και ο κύριος Μπέρμαν. Τις εξορρυκτικές βιομηχανίες. Πρέπει αυτό να μπει στο πρόγραμμα εργασιών στο μέλλον. Είδατε τον πρόσφατο αμερικανικό νόμο, είναι καλό το μοντέλο. Ε, ε θα πρέπει να δώσουμε χρήματα για την βελτίωση του κλίματος, ε, της οικονομίας ε, και την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσεων. Ορισμένες χώρες της Ένωσης δεν πληρώνουν φόρους στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται στον, στις αναπτυσσόμενες χώρες και προτιμούν α, ε, α, ε, τους φορολογικούς παραδείσους. Επίσης, ε, υπάρχει ανάγκη για νέο δημοσιονομικό μέσο που θα αντικαταστήσει την, το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας και θα χρειαστεί και ε, παγκόσμια πρόσβαση στην καθαρή ενέργεια. Είναι σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη, αναπτυξιακή βοήθεια και έτσι θα βελτιωθεί ε, το κλίμα. Συγχαρητήρια με αυτά, για αυτά που κάνετε μέχρι τώρα. Δεν έκανα τόσο ερωτήσεις όσο σημαντικά θέματα όπως ας πούμε βοήθεια για τη αποτελεσματικά μέτρα για το εμπόριο γιατί είναι σημαντικό ο ρόλος που μπορούμε να παίξουμε στις χώρες εκτός Ένωσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ωφέλη για τα κράτη-μέλη μέσα από αυτές τις πολιτικές. Σας κατευχαριστώ και τώρα θα μιλήσω κι εγώ Κύριε Πίμπαλξ, όλο και περισσότερο παρατηρούμε εμείς οι πολιτικοί ότι οι πολίτες είναι πολύ περήφανοι για αυτά που κάνει η Ένωση ως προς τη βοήθεια, την αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν καταλαβαίνουν όμως γιατί δεν είμαστε πιο απαιτητικοί, γιατί δεν βάζουμε περισσότερους όρους. Μπορεί μερικές χώρες να το θεωρούν αυτό ουτοπικό για, για μερικές χώρες αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να είμαστε πιο απαιτητικοί με χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προηγουμένως όταν μιλούσατε κατάλαβα ότι άκουσα ότι θέλετε να ενδυναμωθεί το σύστημα, να υπάρξουν περισσότεροι όροι. Η κυρία Σαργεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίμπαλγκς, σήμερα ξανασυζητούμε την έκθεση, την αξιολογική έκθεση και εκεί γίνεται λόγος για την συμπεριληπτική ανάπτυξη. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς πώς τη βλέπετε αυτή την έννοια, γιατί και εγώ και ο εισηγητής ο κύριος Κάσμαν θα μπορούσαμε να βοηθηθούμε πολύ από αυτά που θα μας πείτε. Έπειτα, το θέμα των εμπορευμάτων, η Κομισιόν ανέλαβε την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες που παίζουν μεγάλο ρόλο στις σχέσεις μας με την Αφρική. Εσείς και η γενική σας διεύθυνση τι ρόλο παίζετε για τις πρώτες ύλες, την πρωτοβουλία των πρώτων ύλων. διότι γενικά ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος Δεχόχτα από την εσωτερική αγορά και το διεθνές εμπόριο ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εσείς τι φρονείτε. Μετά το θέμα των οικοπεδοφάγων. Εσείς πώς το βλέπετε, ή υπάρχει ενωσιακή ευθύνη για το θέμα αυτό στην Αφρική, της οικοπεδοφαγίας στην Αφρική. Ή άμα δεν το πω οικοπεδοφαγία, ας πω ανέβρεση νέων γεών από αναπτυσσόμενες χώρες με τρόπο για καλλιέργειες που δεν ωφελούν απαραίτητο στον πληθυσμό. Και νομίζω μια άλλη καινούργια έννοια είναι και η θαλασσοφαγία. Δηλαδή το γεγονός ότι Ευρωπαίοι ψαράδες εκμεταλλεύονται θαλάσσιες περιοχές στη, κοντά στις δυτικές ακτές της Αφρικής και έτσι εμποδίζουν τους τοπικούς ψαράδες να κερδίσουν τη ζωή τους. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για τη θαλασσοφαγία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τεκάιζερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φυσικά συμφωνώ με τα ερωτήματα που θέτει η ομάδα μου, ιδιαίτερα ως προς μια νομοθετική πρωτοβουλία για τα ορυχεία, για τις εξορρυκτικές δραστηριότητες, αλλά δεν θα επιμείνω γιατί το ανέφεραν και άλλοι. Εγώ θα ήθελα κύριε Πίμπαλγκ να γνωρίζω τα εξή, Να γίνει μια ανακοίνωση της Κομισιόν για την κοινωνική προστασία όπως το, είχε, το είχαν προτείνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2007 αν δεν απατώμε. Νομίζω ότι θα ήταν διπλά καλό αυτό γιατί καταρχάς σε ένα ψήφισμα της Επιτροπής μας που είναι κρίθη από την Ολομέλεια για την υγεία στην Υποσαχάρη Αφρική είχαμε μιλήσει για τη σημασία που έχει η ανάπτυξη ασφαλιστικών οργανισμών στην Αφρική ή συμπληρωματικών πέρα από την βασική ασφάλιση. Τώρα όμως με βάση τις εξελίξεις που παρατηρούνται στη Βόρεια Αφρική φαίνεται ότι τα διεφθαρμένα και αυταρχικά καθεστώτα που δεν μπορούμε λόγω εν ονόματι της μη παρέμβασης δεν μπορούμε να τα ρίξουμε και αυτό είναι φυσικό θα μπορούσαμε τουλάχιστον στις χώρες αυτές να ζητήσουμε κάποια αρρωγή της κοινωνίας των πολιτών που μπορεί να αποδειχτεί πολύ σημαντική στο μέλλον. Σήμερα είναι διπλό το συμφέρον που θα είχαμε να εξυπηρετήσουμε και την υγεία αλλά και τη διατήρηση μιας κοινωνίας των πολιτών κινημάτων που βλέπουμε να γεννιούνται παντού στην Αφρική και να τα καταστήσουμε εχμήν του δόρατος της νέας μας στρατηγικής. Στη βράση κολλάει το σίδηρο κύριε, κύριε Επίτροπε. Θα έπρεπε νομίζω λοιπόν αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι παραπάνω για την κοινωνική προστασία, για τις κοινωνικές ασφαλίσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτρόπε, δεν θα... δεν θα επαναλάβω αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι και με τα πλήστα, με τα πλήστα εξ αυτών συμφωνώ. Άλλωστε έχουμε καθορίσει πολιτικές αρκετές φορές με πολύ σωστά και δυνατά ψηφίσματα. Θα εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου, ενός πολύ μικρού κράτους, το οποίο με τόσα πολλά προβλήματα καταφέρνει να διαχειρίζεται σωστά την αναπτυξιακή βοήθεια και να είναι πρωτοπόρο θα έλεγα και να εκφράσω και την προσωπική μου περηφάνεια για την εμπλοκή μου σε αυτή την προσπάθεια, την προσωπική μου εμπλοκή και την συμμετοχή. Ωστόσο κύριε Επίτροπε θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς κρίνετε την πεισματική άρνηση της Τουρκίας να αποδεχθεί ή να προσκαλέσει την Κύπρο στην, σύνοδο, στην τέταρτη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη τον άλλο μήνα. Εσείς θα εκπροσωπείτε τους 26 όταν θα πάτε εκεί. Η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πού βρίσκεται. Δηλαδή είναι δυνατόν να αποδεχτούμε μια χώρα πρωτοπόρο στην αναπτυξιακή βοήθεια να μην την δέχονται καν να συμμετάσχει σε μια σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Crétu, c'est à vous. Thank you very much, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που ήρθε να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Πολιτικής για τον επόμενο χρόνο. Με λύπη άκουσα ότι από τα νέα κράτη-μέλη μόνο η Κύπρος πληρεί τους αναπτυξιακούς στόχους. Δεν θα μπορούσαμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη με κάποιο τρόπο να ε, ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ας πούμε κινητοποίηση της κοινή γνώμης στα κράτη-μέλη Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό θα είναι αποτελεσματικό. Τουλάχιστον στη δική μου τη χώρα είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε τον κόσμο ότι θα πρέπει να αναλάβουν υποχρεώσεις για άλλους, προς άλλους λαούς. Όχι μόνο επειδή, όχι επειδή η κοινή γνώμη είναι εγωιστική, αλλά πολλές φορές και η πολιτική είναι λαϊκιστική. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος τρόπος άλλος ώστε να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν. Επίσης, ένα άλλο θέμα, πώς θα ε, βεβαιωθούμε ότι όχι μόνο θα γίνει η φωνή μας ακουστή, αλλά ε, και σεβαστή από τη διεθνή κοινότητα. Έχουμε τώρα την Σύνοδο Κορυφής στην Κωνσταντινούπολη και την, επόμενη, την ε, περασμένη εβδομάδα περάσαμε αυτό το ψήφισμα με πολλές συστάσεις από τη δική μας την πλευρά. Και γενικά εκδίδομαι πολλές νομοθετικές πράξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διάφορα διεθνή θέματα, χωρίς να είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι οι πρωτοβουλίες μας λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα τώρα με τα Ηνωμένα Έθνη και το καθεστώς μας του παρατηρηθεί, πώς θα δώσουμε συνέχεια στις ιδέες που εκφράζονται σε όλα αυτά τα ψηφίσματα. Πώς θα βεβαιωθούμε ότι θα λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόγκα έχει το λόγο. Merci, Monsieur le Commissaire. Euh, je voudrais vous, vous interroger sur la question. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τα PTON. Μιλήσατε για τον ειρηνικό, για τις ε, προτεραιότητες τον ειρηνικό και την Καραϊβική. La, la proposition θα ήθελα να μας μιλήσετε για το μελλοντικό ε, πλαίσιο σύνδεσης. Μιλήσαμε στη Νουμέα για τη σύνδεση με τα ΠΤΟΕΝ. Ναι. Για τα ε, υπερπόντια εδάφη. Ναι και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η πρότασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε. Μας ε, διευκρινίσατε ότι έχετε πολλά εργοτάξια και στη Βόρεια Αφρική και στην ακτή Ελεφαντοστού και Υπάρχουν και άλλες προτάσεις από τους ευρωβουλευτές. Είναι Ηράκλειο το έργο σας, γιατί η χρηματοδότηση, χαιρετίζω αυτά που είπατε, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις στα κράτη-μέλη για να επιτύχουν το στόχο του 0,7% και νομίζω ότι σε, με βάση την αρχή του shame and blame θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Η Πορτογαλία που έχει τόσο μεγάλη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ε, ανταποκρίνεται, ενώ πλουσιότερα κράτη όχι. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είχαμε τον ε, Επίτροπο για τη Διεύρυνση, κύριο Φίλε. Πολλά κεφάλαια πρέπει να ε, ανοίξουν ακόμα. Όταν διαπραγματευόμαστε με νέα κράτη-μέλη πρέπει να τους ε, καταστήσουμε σαφές ότι γρήγορα θα κληθούν και στην αναπτυξιακή βοήθεια να επιδιώξουν το ευρωπαϊκό επίπεδο. Να βάλουμε στη συζήτηση 0,7%. Εντάξει, δεν θα είναι κριτήριο για την προσχώρηση, την ένταξη, αλλά παντού πρέπει να τονίζουμε και να προωθούμε αυτό το στόχο που πρέπει να πετύχουμε. Είμαι περήφανος διότι η Κομισιόν και η Επιτροπή από κοινού το Μάιο στη Βουδαπέστη θα ολοκληρώσουν τον διαρθρωμένο διάλογο και οι τοπικές αρχές, η κοινωνία των πολιτών θα ενισχυθούν. Αυτό είναι μια αναπτυξιακή βοήθεια που πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερο για να κάνουμε καλύτερη, καλύτερο κυβερνητικό έργο να έχουμε. Πώς θα το πετύχουμε. Θα φροντίσουμε για τα κοινωνικά συστήματα ε, ασφάλειας, ασφάλισης, ε, παιδείας ε, το Κόγκο είναι μια χώρα που δεν έχει ε, φορολογικά έσοδα γιατί δεν υφίσταται ένα σύστημα που θα μπορεί να εισπράττει τους φόρους εκεί. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επίσης, οι χώρες κατοφλίου, οι αναδυόμενες οικονομίες. Αν δούμε το στόχο της χιλιετίας, για παράδειγμα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τη θνησιμότητα των ε, παιδιών και γυναικών. Αν δούμε ότι οι θάνατοι εδώ στην Ινδία είναι περισσότεροι από ό,τι σε ολόκληρη την Ποσαχάρη Αφρική, ε, δεν μπορούμε αυτό να το επιτρέψουμε. Ε, αναπτυξιακή βοήθεια σε, ένα, σε μια χώρα στην Ινδία, εντάξει την υποστηρίζω, αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει πυρηνικά όπλα και έχει το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα διαστημικό, διαστημικών ερευνών. Άρα λοιπόν υπάρχει περιθώριο για άσκηση πιέσεων στην ελίτ αυτή τη χώρας. Τώρα, για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, εδώ υπάρχουν πολλές ε, ιδέες για το πώς θα χρησιμοποιηθούν. Είναι περίπλοκος ο φόρος αυτός έτσι όπως ονομάζεται. Μπορούμε να τον ονομάσουμε φόρο κατά της φτώχειας, γιατί έτσι θα γίνει κατανοητό πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους φόρους αυτούς και πώς τα έσοδα αυτά θα ε, ε, καταναλωθούν και θα δοθούν για ανάπτυξη στο μέλλον. Επίσης είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση σήμερα το πρωί για την σύγχυση των ρόλων μεταξύ ανθρωπιστικών και στρατιωτικών φορέων, ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Βλέπω εδώ μια τάση, για αναπτυξιακή πολιτική, ανθρωπιστική βοήθεια να υποτάσσεται στις στρατιωτικές επιλογές. Πρέπει όλοι να φροντίσουμε η ανθρωπιστική βοήθεια να, διαχω... να παραμείνει αυστηρά διαχωρισμένη από τη... τις στρατιωτικές δράσεις. Τελειώσαμε. Α. Θα ήθελα τώρα να είσαστε ιδιαίτερα σύντομοι γιατί μιλήσατε και πριν. Μιλώ εκ μέρους του κυρίου Κέλλερ που είναι στην Ινδία και θέλει να κάνουμε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Δηλαδή, τι θα κάνετε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές και την αρχιτεκτονική των δημοσιονομικών μέσων, μηχανισμών, πώς θα μεταρρυθμιστεί το DCI, το μηχανισμό της Αναπτυξιακής Συνεργασίας και τι έχετε υπόψη σας εδώ. Ο κύριος Πίμπαλξ, για να απαντήσει. Καλό κουράγιο να απαντήσετε σε όλα αυτά. Κοιτάξτε, θα αρχίσω λέγοντας ότι η αναπτυξιακή συνεργασία είναι πιστεύω το πιο πολύπλοκο, πιο πολύπλοκος τομέας πολιτικής που μπορεί κανείς να βρει στην Ένωση γιατί πρέπει να απαντήσει να ανταποκριθεί σε πολλές ανάγκες και προβλήματα και δεν είναι πάντα σε θέση να δίνει ικανοποιητικέ απαντήσεις για όλους τουλάχιστον. Θα προσπαθήσω πάντως να απαντήσω τουλάχιστον σε ορισμένες από τις ερωτήσεις και στους υπόλοιπους να δώσω μερικές απλώς ιδέες. Το ερώτημα για το ότι δεν υπάρχει επαρκής συντονισμός και κατανομή εργασίας μεταξύ των 27. Αυτό βελτιώνεται. Όπως ας πούμε με την IT, με την ακτή του Ελεφαντοστού και με τον Νότιο Σουδάν. Εκεί νομίζω θα φανεί ότι έχει βελτιωθεί ο συντονισμός, αλλά για να μεταφερθούν όλα όσα χρειαζόμαστε να μεταφέρουμε εκεί και γρήγορα θα χρειαστεί πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Πρέπει να γνωρίζουμε κάθε φορά τι ακριβώς, σε τι ακριβώς επίπεδο βρίσκονται οι, θέσεις, οι σχέσεις μας με κάθε χώρα. Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις μεταξύ και συνεννοήσεις μεταξύ γενικών διευθυντών. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε να σπαταληθούν χρήματα Το θέμα δεν είναι πρόβλημα εθνικής κυριαρχίας αλλά υπεύθυνη χρήσης των κονδυλίων. Μπορεί στο μέλλον να ζητήσουμε διαχείρισή τους με πιο με διαφορετικό τρόπο όπως κοινούς προγραμματικούς κύκλους και τέτοια για να μην χαθούν τα 6 δισεκατομμύρια. Πρέπει επίσης να αναλύσουμε όσο δυνατόν περισσότερο το θέμα της, του εξυγχρονισμού αλλά θα συζητήσω και με το προσωπικό μου τι άλλο μπορεί να γίνει για να δούμε τι, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για θέματα πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας, διότι υπάρχει όντως πολύ λίγη πρόοδος επ' αυτού και δεν πρόκειται να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις αν δεν λυθεί αυτό το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάντως θα κάνουμε την προσπάθεια για τα επιστημονικά προγράμματα. Θα έπρεπε πράγματι να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Αν και μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας δεν πρόκειται για υψηλά ποσά. Αλλά προσπαθούμε να προωθήσουμε και επιστημονικά προγράμματα με επιστημονικά στοιχεία για την ανάπτυξη της κάθε χώρας. θα στείλουμε κείμενο σχετικό εν καιρό το θέοντι. Για θέματα διαφάνειας συνεννοήθηκα με τον Επίτροπο Μπαρνιέ πριν από μερικές εβδομάδες και υποστηρίζει και αυτό την ίδια προσέγγιση. Τον, το φθινόπωρο θα κάνουμε προτάσεις για πλήρη ή πληρέστερη διαφάνεια. Εγώ δεν είδα καμία αντίφαση μεταξύ των προθέσεων του και των δικών μας. Θα έλεγα μάλιστα ότι είμαι διατεθειμένος να ξαναέρθω αν δεν έρθει εκείνος να σας εξηγήσω το κοινό μας, την κοινή μας αντιμετώπιση. Αυτό είναι υπόσχεση. Για μένα ναι. Γιατί είμαι υπεύθυνο και εμένα να ρωτάτε άμα δείτε ότι τίποτα πάει στραβά. Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, νομίζω ότι θα έρθει. Γιατί υπάρχει μια σωστή θετική δυναμική μεταξύ μας μέχρι τώρα. Πρόεδρε, πρόεδρε, ζητώ αποσαφήνιση. Σαφήνιση. Ευχαριστώ. Όχι τώρα, όχι τώρα. Α, όχι τώρα, καλά. Το επεξεργαζόμαστε λοιπόν, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτε παραπάνω μέχρι να γίνει η αξιολόγηση. Παρακαλώ πρόεδρε, παρακαλώ γιατί εδώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Μπορώ να ζητήσω αποσαφήνιση. Μα να διακόπτεται τον επίτροπο, τι πράγματα είναι αυτά. Κοιτάξτε, είπατε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να υπάρξουν προτάσεις και για τον Dot Frank. Έχω ρωτήσει και εγώ τον Μπαρνιέ και εδώ τίθενται δύο θέματα. Το ένα είναι η διαφάνεια και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Το άλλο όμως είναι το θέμα της υπευθυνότητας. Μπορείτε να του ζητήσετε, να τον ρωτήσετε αν θα τα συνδυάσει διότι Νομίζω ότι θα δώσει το βάρος στο ένα από τα δύο θέματα. Το λαμβάνω υπόψη αυτό. Έχετε δίκιο, δεν δουλεύει πάνω στα θέματα ε, συγκρούσεων. Μέχρι τώρα λειτουργούσαμε με βάση τις εκθέσεις αναχώρα. Εγώ υπόσχομαι να το δω αυτό. Τώρα, γιατί μια φωνή ε, συμμετείχα σε μια δημόσια συζήτηση και κάποιος είπε έχουμε πολλές φωνές και δεν έχουμε μήνυμα. Είπα δεν είναι τόσο κακό αυτό, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε μεγάλη υποστήριξη ε, ώστε να βελτιώσουμε και τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και να ε, ε, προβάλλουμε ένα μήνυμα. Πρέπει λοιπόν και να βοηθήσουμε την υπάτη εκπρόσωπο στην ανάπτυξη της συνεργασίας. Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες λεπτομέρειες που θα βελτιωθούν οι εξωτερικές σχέσεις ε, θα πρέπει να βελτιωθούν ούτως ώστε να επιτύχουμε να μιλάμε με μια φωνή. Για την ερώτηση του Charles για τον παιδαγωγικό ρόλο. Εγώ θα ήθελα σε οποιαδήποτε συζήτηση και επιτροπή να θέτουμε το θέμα αυτό. Βεβαίως είναι σημαντικό όταν έχουμε ε, στήριξη του προϋπολογισμού να εξηγούμε τα ωφέλη, τους κινδύνους αλλά και τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου και στο μέλλον για την καινοτομία και τη συνένεση του Washington στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να δούμε καλύτερα τις πολιτικές ε, για την ανάπτυξη. Υπάρχουν χώρες που πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Καμιά φορά χρειάζονται και ανορθόδοξοι τρόποι για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα ε, και για τις καινοτομίες ε, ε, να αξιοποιήσουμε την επιστημονική κοινότητα δηλαδή. Τώρα τις 27 πολιτικές και τη μία πολιτική. Νομίζω ότι η δημοσιονομική υποστήριξη είναι σημαντική. Αν γίνει κατανοητή και εφαρμοστεί η δημοσιονομική υποστήριξη, αυτό θα είναι μεγάλο βήμα. Και μετά θα έχουμε εθνικές στρατηγικές, ε, τις εκθέσεις τους. Όταν ε, ε, επισκεπτόμεθα και μιλάμε με τις χώρες μέλη, δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις στις προσεγγίσεις. Αλλά όταν πρόκειται στο διατάφτα δημιουργούνται προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή. Δεν αντιπαλεύουμε ο ένας τον άλλον ούτε στο Συμβούλιο, αλλά πολλές φορές ε, ε, παρουσιάζεται στα δημοσιεύματα μια διαφορετική εικόνα. Αυτό είναι μια πρόκληση. Τώρα για τον επιχειρηματικό τομέα. Ε, εγώ θέλω να δω καλύτερα το θέμα αυτό. Πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα για να επισημοποιηθεί, αν θέλετε, ένα κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου. Ε, τώρα για την ανάπτυξη χωρίς ε, αποκλισμούς στο βαθμό που δεν ε, υπάρχουν στοιχεία δεν, και δεν είναι επίσημα τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και η δομή της νέας Γενικής, Διεύθυν, Γενικής ΕΚΟ θα βελτιώσει τη λειτουργία της. Ε, βέβαια... Ε, ε, δεν μπορώ να ε, σχολιάσω από τώρα το περιεχόμενο της έκθεσης. Θα πρέπει να δούμε λεπτομερέστερα το θέμα και να υποβάλλουμε προτάσεις και για τις καινοτομίες και για την καλύτερη δημοσιονομική πλευρά. Θα, θα γίνει ανάλυση επιπτώσεων και θα επανέλθουμε. Ε. για τη διατροφή, ασφάλεια τροφίμων, ε, κερδοσκοπίες. Στηρίζομαι την ε, Γαλλική Προεδρία και τις δραστηριότητες στην G20 προσπαθούν να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό και νομίζω ότι μπορεί να έχει μια περιορισμένη επιτυχία. Αν δούμε τι γίνεται επί τόπου και μάλιστα εμείς αλλάξαμε τις πολιτικές μας ε, και στη Γεωργία και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η κατάσταση είναι καλύτερη τώρα από ότι το 2008. Δεν πρέπει να είμαστε αυτάρεσκοι σε σχέση με αυτά που κάναμε για την επισητιστική ασφάλεια, αλλά σίγουρα η κατάσταση βελτιώθηκε. Και ένας λόγος που είχαμε, είχαμε ένα δισεκατομμύριο για την πρωτοβουλία για την επισητιστική βοήθεια και είχαν και καλή συγκομιτή σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι αν ενισχύσουμε την προσέγγιση μας για μια βιώσιμη, ένα βιώσιμο γεωργικό τομέα, εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, ώστε να μπορούν να έχουν αυτάρκεια επισητιστική οι χώρες αυτές. Σε αυτό το στάδιο θα έλεγα ότι οι εκθέσεις που λαμβάνω δεν είναι ανησυχητικέ, αλλά απαιτούν πολύ προσοχή στο μέλλον για την κοινωνική ρήτρα. Θα επανέλθω αργότερα. Και θα απαντήσω για την ερώτηση του Μάικ. Είμαι ευγνώμων για τα καλά σου λόγια καταρχήν. Τώρα για τα βασικά που έθεσες, για τις θεμελιώδεις αξίες Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές μας προβοκάρουν επίτηδες, χωρίς η, γνώμη, η κοινή γνώμη των χωρών αυτό να συμφωνεί. Γι' αυτό δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα της προβοκάτσιας. Σίγουρα όμως δεν θα πρέπει να δίνουμε ε, χρήματα όταν παραβιάζονται τέτοιες αξίες. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις χώρες εταίρους. Ε, το σημαντικό είναι να έχουμε συνεπή πολιτική. Θέλω συνεπή προσέγγιση στη δημοσιονομική στήριξη. Θα λάβουμε υπόψη μας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και θα, είμαστε, θα κινηθούμε όλοι μαζί. Είναι σαφές ότι πρέπει να δράσουμε με μια φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πρέπει να επιτρέπουμε υπαναχωρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν λέω να αποσύρωμε την βοήθεια, αλλά το συγκεκριμένο μηχανισμό τη βοήθεια. Δεν θα τιμωρήσω με το λαό αυτών των χωρών, αλλά δεν μπορούμε να συνεργαζόμεθα με τι κυβερνήσει του όταν έχουμε θεμελιώδει διαφωνίε και όταν βλέπουμε ότι αυτοί υπαναχωρούν. Συμφωνώ λοιπόν με αυτή την προσέγγιση. Χρειάζεται λίγη υπομονή και από εσάς και μια συντονισμένη προσέγγιση και για το Παγκόσμιο Ταμείο ισχύει αυτό. Θα πρέπει να μην παρεκκλίνουμε και να μην υπάρχουν διαφορετικές ε, παρουσιάσεις προς τα έξω. Πρώτα να συζητούμε και να ενεργούμε σύντομα. Ε, ενώ τώρα ε, σπέβδουν όλοι να ε, πάρουν θέση, πράγμα που δημιουργεί μεγάλη αμηχανία και δύσκολη θέση σε άλλους. Για τα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί θα υποστήριζα μάλλον τους εταίρους μας. Νομίζω ότι η ψηφοφορία που χάσαμε έδειξε καλά ότι θα έπρεπε να είχαμε δουλέψει σκληρότερα και το κάνουμε τώρα αυτό. Ε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και εγώ δουλέψαμε για να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το θέμα. Αλλάξαμε λίγο την ταυτότητά μας, αλλά είμαστε ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε στα Ηνωμένα Έθνη ως παρατηρητές. Δεν ζητάμε και τόσα πολλά. Δώσαμε τις εξηγήσει και είπαμε, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ε, δώσαμε τις εξηγήσει. Είπαμε ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, είπαμε ότι είναι σημαντικό και ελπίζω ε, στο μέλλον οι χώρες εκεί να μας υποστηρίξουν. Αν δεν το κάνουν, τότε φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται για τους εταίρους τους. Ας μην κρίνουμε με βάση το παρελθόν. Εμείς πήραμε το μάθημά μας και πραγματικά δόθηκαν πολλές εξηγήσεις. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν εξηγήσαμε τη σημασία της ψηφοφορία για μας και το κάναμε σε όλα τα επίπεδα, στι νοιέ, στις κυβερνήσεις, σε ανώτατο επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι παραμελήσαμε ούτε και τη μικρότερη χώρα μέσα στα Ηνωμένα Έθνη. Απευθυνθήκαμε σε όλες τις χώρες και στο μέλλον οι ψηφοφορίες θα δείξουν ποιος θέλει να συνεργαστεί και ποιος δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ. Δεν λέω, ε, είναι ακόμα ελεύθερη ψήφο. Η κάθε χώρα, ε, ψήφος κατά συνείδηση δηλαδή, η κάθε χώρα έχει την άποψή της. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι εταίροι μας ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις μας και πρέπει και εμείς ε, να ζητήσουμε τη θετική ψήφο, να εξηγούμε ξανά και ξανά. Πολλές φορές είναι λεπτά τα θέματα, όπως μας λένε, γιατί ε, υιοθετήσατε τη συνθήκη της Λισαβόνα κλπ. Ε, πάντως δεν πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε για μια θετική ψήφο. Για το 0,7 και αν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Νομίζω ότι αυτό επισέρχεται πολύ στην εθνική κυριαρχία. Πήγα και στη Ρουμανία, μίλησα με την κυβέρνηση και είπαν μέχρι το, μας είπαν μέχρι το 2015 θα τα καταφέρουμε και το είπαν και ήταν τώρα είμαστε στο 2010 μας λέγανε ε, έχουμε πολλές δυσκολίες ε, αργότερα θα τα καταφέρουμε νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, εξετάσεις ε, δηλαδή εκθέσεις από ομοτήμους να μην φανεί ότι πιέζει εξαναγκάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, κινητοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση. Για την εξωτερική βιομηχανία... Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Μπέρμαν. Ε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την πρόταση αυτή από την υπηρεσία μου τώρα. Μιλήσαμε για το, τη στάση μας στα δικαιώματα πνευματικής διοκτησίας και τι σημαίνουν όλα αυτά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα για τα φάρμακα, την πρόσβαση στην υγεία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της ε, συνοχής της πολιτικής στην ε, Επιτροπή δεν υποβάλλουμε προτάσεις σε αυτό το στάδιο. Πάντως κάθε βήμα μας πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Για την ε, ερώτηση της Προέδρου για τους όρους, ε, δηλαδή την έννοια της αιρεσιμότητας, αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ γιατί σε τελευταία ανάλυση Μιλάμε για τα χρήματα των φορολογουμένων, για την αξιοπιστία μας. Μπορούμε να συζητούμε ειλικρινά, ανοιχτά με τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και προς τον εαυτό μας και προς τους εταίρους μας. Η κυρία Σαρτζεντίνη, τι είναι η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Δεν θα αποπειραθώ ορισμό αν υπάρχει ανάπτυξη, αν δημιουργείται πλούτος, θα πρέπει μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες να διανέμεται ε, ισότιμα. Να έχω δηλαδή κοινωνικά συστήματα που θα κατανέμουν τα εισοδήματα πιο ισότιμα στον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι δηλαδή κατεξοχήν αύξηση του ΑΕΠ, αλλά πώς γίνεται η δίκαιη ανακατανομή σε όλη την κοινωνία. Για την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε, νομίζω ότι δεν ήταν και τόσο άσχημα το κείμενο, η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε. εντάχθηκε στην πολιτική συνοχής για την ανάπτυξη. <laughs> Τώρα, για την ρουσικοπεδοφάγου στην παράνομη ε, κατοχή γης ε, στη Σαουδική Αραβία. Ε, είναι οι εταιρείε από τη Σαουδική Αραβία, Κίνα, Ινδία που παίζουν ρόλο εδώ. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα είναι η πλήρης διαφάνεια και η δημοσίευση των τίτλων ιδιοκτησίας και της αλλαγές. Πολλές φορές μας λένε ότι βάζουμε πολλούς όρους ε, και προϋποθέσεις και δεν καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα. Όμως μόνο με διαφάνεια θα πρέπει ή ε, τα συμβόλαια να ε, δημοσιεύονται, να είναι διαφανή για να ξέρουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Γιατί η Βερονίκ Τεκάιζερ δεσμεύομαι να εργαστώ για την ανακοίνωση για το 2012 και για το 2007 έγινε, είναι ένα οριζόντιο θέμα σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε για την ε, ανακοίνωση για το 2012. Κυρία Θεοχάρους, πολύ εκτιμώ αυτά που κάνετε στην Κύπρο και αυτό με κάνει να ελπίζω ότι οι χώρες που εντάχθηκαν μετά το 2004 θα ακολουθήσουν. Υπάρχει ηγεσία εδώ όχι μόνο ε, σε χαμηλό αλλά και σε ανώτερο επίπεδο για την Κωνσταντινούπολη ε, στα Ηνωμένα Έθνη πιστεύω ότι θα πρέπει να συμμετέχετε. Δεν το γνώριζα. Είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην λάβει πρόσκληση στα Ηνωμένα Έθνη. Εκπλήσωμαι που το ακούω, δεν το ήξερα και θα το δούμε το θέμα αυτό. Και η αντιπροσωπεία της Ένωσης, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να δει ποια είναι αυτά τα θέματα που αφορούν την δίκαιη μεταχείριση των αντιπροσωπιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα φροντίσω το θέμα αυτό της συμμετοχής σας, της συμμετοχής ε, όλων των κρατών μελών άλλωστε. Ελπίζω να ε, συμβεί αυτό. Για την κυρία Κρετού και τις συστάσεις Ήμουν στο Ουσμπεκιστάν δυστυχώς και δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στη συζητήση στο Κοινοβούλιο και λυπάμαι που η έκθεση δείχνει ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν λαμβάνονται παρκώς υπόψη οι απόψεις του. Θα το βελτιώσουμε αυτό το θέμα. Αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Θα λάβουμε υπόψη μας τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές δεν ταυτίζονται οι απόψεις μας, αλλά θα φροντίζομαι να εισακούονται οι απόψεις σας και δεν νομίζω για τα θέματα αυτά να έχουμε διαφορές απόψεις. Για τον κύριο Πόγκα ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό των υπερποντίων εδαφών και χωρών. Θα είμαστε ε, προετοιμασμένοι και σε αυτό το στάδιο ε, έχουμε εντοπίσει κάποιες δυσκολίες όπως το μέγεθος είναι πολύ μικρές οι χώρες αυτές και τα εδάφη. Είναι όμως ε, χώρες ε, εδάφη κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να διατηρήσουν αυτό το καθεστώς, οπότε πρέπει να μας απασχολήσουν τα προβλήματά τους. Για την ερώτηση του κυρίου Νόιζερ, Έχουμε μια εξαιρετική πρόκληση να αντιμετωπίσουμε, αυτό φαίνεται και εδώ, εν προκειμένου, με τις εξελίξεις στη Βόρειο Αφρική ειδικότερα. Θα έλεγα ότι πάντα πρέπει να φροντίζομαι ε, για την ισορροπία των σχέσεων που υπάρχουν ε, και πολλές φτωχές χώρες στην περιοχή. Μιλάμε για τη Βόρειο Αφρική ξεχνώντας ότι υπάρχουν απελπιστικές συνθήκες σε άλλες χώρες. Οι νέες προκλήσεις δείχνουν ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις πιο φτωχές χώρες. Βεβαίω αναγνωρίζω τα προβλήματα στη Βόρειο Αφρική, αλλά δεν είναι τόσο θέμα αναπτυξιακή βοήθεια εδώ, ή είναι θέμα υποστήριξη, διακυβέρνηση και τέτοια θέματα. Θεμητό και σωστό να βοηθηθούν οι χώρε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα βήμα παραπέρα έχουμε τη Σαχάρα, την υποσαχάρια περιοχή που εκεί πεθαίνει κόσμος από αρρώστιες, υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Ε, Συν το χρόνο ίσως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κεκτημένο για την αναπτυξιακή συνεργασία Τώρα, πρέπει να αρχίσουμε από τα πιο, τις πιο ευάλωτες χώρες, λιγότερο αναπτυγμένες και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. για χώρες όπως την Ινδία ε, θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται τόσο. Όχι, θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν και να βοηθούν τα κράτη-μέλη ίσως, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στοχεύει τους πιο ευάλωτους ε, η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία πάντοτε θα έχουν θυλάκους ένδυας, αλλά θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά μέσα από ε, διμερείς σχέσεις ή φιλανθρωπικές κινήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους. Τώρα γιατί το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να βοηθηθούμε και από την G20 για την επιτυχία. Ε, πρέπει επίσης να δούμε πώς θα απαντήσουμε αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. <laughs> Για η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά δεν ε, παρέχει στρατιωτική υποστήριξη, παρέχουμε ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Η ακτή του αλεφαντοστού είναι ένα καλό παράδειγμα, αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν συνηθίζαμε να συνδέουμε ή να συζητούμε άλλες μορφές βοήθειας. Δεν είναι αυτή η πρακτική μας. Ίσως κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω ότι και εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς εστιάζουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, όχι τη στρατιωτική. Ούτε τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές, γιατί τέλεισε και ο χρόνος. Ε, μίλησα στην Επιτροπή Σούρε, παρουσίασα τις απόψεις μου, δεν προλαβαίνω να το πιάσω αυτό τώρα το θέμα, πάντως τώρα στην Επιτροπή θα γίνει γιατί έγιναν και σεμινάρια. Έχουμε τώρα το, τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα εγκρίνουμε μία πρόταση ε, στη συνάντηση 29 και 30 Ιουνίου στην Επιτροπή. Οπότε σε αυτό το στάδιο δεν μπορώ να προσθέσω περισσότερα από αυτά που είπα και στην Επιτροπή Σούρε. Η κυρία Κέλλερ λοιπόν μπορεί να δει τι είπα εκεί. Just to mention, Commissioner... Κύριε έρχεστε πιο συχνά στην Επιτροπή μας από ό,τι πολλοί συνάδελφοι και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερος. παρακαλώ. Σε λίγο θα αρχίσουμε τις ψηφοφορίες και γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε λίγο ησυχότεροι όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν τώρα. Βγάλτε τις κάρτες σας. Σήμερα όλα θα τα κάνουμε ηλεκτρονικά. 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing, testing. Παρακαλώ. Αντσι, μπράβο. Λοιπόν, αρχίζουν οι ψηφοφορίες. Έχουμε 15 λεπτά. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Να αρχίσουμε τότε. Έχω και εγώ την κάρτα μου. Ωραία. Πρώτα μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν όλοι. Ούτε όλες. Ευτυχώς που είναι δοκιμή, ε. Δουλεύει. Λείπουν λοιπόν, έξι. Πέντε. Έξι πάλι. Όχι, τώρα δύο. Μήπως να αλλάξετε θέση. Αλλάξτε θέση. Σε καμία θέση δεν δουλεύει κυρία Πρόεδρε. Πάλι λοιπόν δύο. Ακόμη. Δεν δουλεύει. Ένας. Α, η Βερονίκ. Τη Βερονίκ περιμέναμε. Ένας λείπει ακόμη, ένας λείπει. Η μία. Α, τώρα είναι όλοι παρόντες. Μην κουνιέται κανείς λοιπόν. Έληξε ψηφοφορία. Να, ορίστε. Λοιπόν, αρχίζουμε. Κρήτον Αρσένης. Τροπολογία 1. Υπέρ... Όχι, όχι, μάλλον είπαμε ηλεκτρονικά ότι θα το κάνουμε. Ηλεκτρονικά είπαμε. Έτσι είχαμε πει. Ε, μου είπατε όλα ηλεκτρονικά. Όχι, τώρα μου λένε όχι όλα ηλεκτρονικά. Λοιπόν, τώρα διανατάσεως της χειρός. Υπέρ. Κα... Ε, μετράτε, μέτρησε κανείς. Κατά. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Α, το φανταζόμουν. Λοιπόν, λοιπόν, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ ανατάσεως. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιο κινητό θορυβεί παρακαλώ κλείστε του, λέει η πρόεδρος. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά την εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 που αντικαθιστά όχι είναι σε τρία τμήματα μάλλον σε τρία τμήματα δεν είναι ναι λοιπόν πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 Α, όχι, περνάμε κατευθείαν στην τροπολογία 13. Υπέρ της 13. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλα, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Πάλι κοντά είναι επαλήθευση, επαλήθευση. Νομίζω ότι απερίφθη, επαληθεύουμε, όμως άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται με διαφορά μίας ψήφου. Τροπολογία... Προφορική τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. τροπολογία 28 υπέρ. Α, όχι, με συγχωρείτε, 25 λέει η 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Έληξε. Εγκρίνεται. υπολογία 33 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίφθηκε αλλά δεν είμαι βέβαιη θα επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία έληξε η ψηφοφορία απορρίφθηκε 34 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 35 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά χες απορρίπτεται 37 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία έληξε απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Ησυχία παρακαλώ. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ όχι α έχει καταπέσει μάλιστα καταπίπτει ή όχι όχι, δεν καταπίπτει. Λοιπόν, 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχει λήξει. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Επομένως τώρα η προφορική 3 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία, έληξε Σαρανταπέντε υπέρ κατά επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Α, όχι, έχει εκπέσει, έχει εκπέσει, έχει καταπέσει. 48. Προπολογία 48. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Τελευταία ψηφοφορία σύνολο της νομοδότησης. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ.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 Merci de respecter les gens qui veulent terminer la réunion en silence. Ευχαριστώ που σέβεστε τους υπόλοιπους και αποχωρείτε ησύχως. Donc, comme demandé lors de notre dernière réunion, nous, nous avons aujourd'hui un deuxième échange de... Έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψε ως προς την έκθεση Κατσμάρεκ σε σχέση σχέση με την ανάπτυξη που ορίζει τη μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την, την έννοια θα δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος και με τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πίμπαλξ. Έχετε αντίγραφα της έρευνας που έχει γίνει και δίνω το λίγο στον κύριο Κατσμάρεκ για να μας κάνει μια εισαγωγή στο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι έχουμε τη δυνατότητα για άλλη μία φορά να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αντικτύπου της αναπτυξιακής πολιτικής Πολλές μη κυβερνητικέ ήρθαν σε επαφή μαζί μου σε σχέση με την πράσινη βίβλο και χαίρομαι διότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να ε, διευρύνουμε, να συζητήσουμε και να διευρύνουμε. Είχαμε συζητήσει το θέμα της ε, πρόσμιξης, του blending, δηλαδή των διαφόρων τύπων αναπτυξιακής βοήθειας. Όσον αφορά το, την πράσινη βίβλο αφορά ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο μέσα στα πλαίσια άλλων αποφάσεων, δηλαδή το πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο, την δημοσιονομική υποστήριξη, χρηματοδοτικά μέσα και ούτω καθεξής. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τη συζήτηση των δύο προγενέστερων συνεδριάσεων θα σταθώ στα πιο σημαντικά σημεία και θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο μήνυμα θέλουμε να αποστείλουμε προς τα έξω. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει μία επαρκή αναπτυξιακή πολιτική και την πλαισιώνει. Αυτό το πλαίσιο συζητήθηκε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνένωσης για την ανάπτυξη δεύτερον. Έχουμε έναν επαρκή ορισμό των στόχων αυτής της πολιτικής από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα πρέπει να εξαλείψουμε τη φτώχεια ή τουλάχιστον να την περιορίσουμε. Δεν έχει σημασία κατά πόσο αυτό βρίσκεται στο πλαίσιο της συνένεσης ή της συνθήκης. Η ουσία παραμένει η ίδια σε σχέση με την πράσινη βίβλο. Ένα άλλο ζήτημα αφορά το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βρει ένα τρόπο να αυξήσει την αποδοτικότητα αυτής της αναπτυξιακής βοήθειας. Το συζητήσαμε και στα πλαίσια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τις φτωχότερες χώρες. Κατά τη συζήτηση στο Στρασβούργο, ορισμένοι ομιλητές ανέφεραν το ότι τρεις χώρες μέσα σε 40 χρόνια κατάφεραν να σπάσουν αυτό το φράγμα και μιλώ για τις φτωχότερες ε, χώρες, οι οποίες θεωρούνται πλέον χώρες με μία επαρκή ανάπτυξη. Επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουμε ως προς το πώς επιτελείται αυτή η ανάπτυξη, η συμπεριληπτική. Θα πρέπει δηλαδή παράλληλα να εξαλείψουμε τις ανισότητες. Δεν πρόκειται για μία ανάπτυξη αυτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η εξάλληψη των ανισοτήτων. Υπάρχουν και κοινωνικά ζητήματα, καθώς και φορολογικά. Ήρθαμε σε επαφή με τον Bill Gates στο Στρασβούργο και όχι και όσοι συμμετείχαν θα θυμόσαστε τι είπε ως προς το φορολογικό. Είναι πεπισμένος ο Bill Gates ότι σε μερικά χρόνια θα αλλάξουν τόσο οι τεχνολογίες ώστε να μπορέσουμε να εισαγάγουμε αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα σε χώρες που δεν τα διαθέτουν ακόμα. Ε, έτσι θα έχουμε ε, μία δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε τις ε, κοινωνικές πολιτικές των ε, κρατών αυτών. Θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα σύστημα το οποίο συσχετίζει την ανάπτυξη με αυτή την συμπεριληπτική ανάπτυξη όπως την ονομάζουμε και όπως κατονομάζουν και οι συνθήκες. Ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι η χρηματοδότηση της υγείας και της εκπαίδευσης. Εάν αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν, η ανάπτυξη δεν θα είναι συμπεριληπτική. Αυτό είναι απαράβατος όρος έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτή την πτυχή της ανάπτυξης. Δηλαδή η ανάπτυξη θα πρέπει να συσχετίζεται με τη μείωση της φτώχειας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δείκτες που αποτιμούν αυτή την αποτελεσματικότητα. Οι δείκτες δεν θα πρέπει να είναι ασθενείς, δεν πρέπει να είναι αδύναμοι. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την ανθρωπιστική βοήθεια, μιλάμε για το χτίσιμο ενός σχολείου κάπου και αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε ότι η πραγματική αποδοτικότητα θα φανεί μερικά χρόνια μετά, διότι πρώτα θα ε, στεγαστούν οι μαθητές, προσληφθούν οι καθηγητές και μετά θα φανούν τα αποτελέσματα. Πρόκειται για μία για την εισφορά δηλαδή, της, ε, τη συνεισφορά της εκπαίδευσης, η οποία φαίνεται μόνο μετά από μερικά χρόνια. Δεν θα πρέπει να επιθυμούμε βραχυπρόθεσμους στόχους, αλλά μακροπρόθεσμους. Ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω τροπολογίες και εγώ έχω προετοιμάσει μερικές. Δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά δεν έχουμε αρκετό χώρο, γι' αυτό χρησιμοποιούμε και το μηχανισμό των τροπολογιών και αυτό αφορά και εμένα, τον εισηγητή. Σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να αναλύσω και να εντάξω όλες τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Τώρα έχετε το λόγο εσείς, η κυρία Κρέτσου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ τον κύριο Κάσμαρεκ, τον εισηγητή μας, για το σκληρή δουλειά που αφιέρωσε στην έκθεση αυτή είναι πολλές οι προκλήσεις, η χρηματοπιστωτική κρίση, η επιστημιστική ασφάλεια και άλλα κλιματικά προβλήματα κλπ. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτηση, στην Επιτροπή ΝΤΕΒΕ θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Ο υψηλός αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής συνδέεται με την αποτελεσματικότητά της. Πρέπει να δούμε τις ανισότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες και να κάνουμε αποτελεσματικότερη έτσι την πολιτική μας. Όταν μιλάμε για ανισότητες, που είναι μεγάλο πρόβλημα συνήθως στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να αναπτυχθούμε σε κοινωνικό-οικονομική ανισότητα, εμφυλή ανισότητα κλπ. Έκανα στην Επιτροπή ΦΑΜ κάποιες τροπολογίες και λείπουν νομίζω από την έκθεση γιατί η ενδυνάμωση των ε, γυναικών είναι ουσιώδη για να μειωθεί η φτώχεια και να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Ένα άλλο πράγμα που θεωρώ σημαντικό στην έκθεση αυτή είναι να ενθαρρύνουμε την πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, παιδεία, όπως είπατε, που είναι σημαντικές για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, Επίσης, όταν μιλάμε για επενδυτικά προγράμματα και έργα, δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε τις αναπτυσσόμενες να θεσέβονται τα, όλα τα πρότυπα, τα διεθνή, αλλά και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, στα πλαίσια της βοήθειας πρέπει να επικεντρωθούμε στην κατάσταση των γυναικών και να μην ξεχνάμε και τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, να επενδύσουμε στα παιδιά και τους νέους μετά από τη συζήτηση με τον κύριο Πίμπαλξ χαίρομαι που ανακαλύπτω στην έκθεση ότι το θέμα της αναπτυξιακής εκπαίδευσης και της ε, ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη το έχετε συμπεριλάβει είναι σημαντικό διότι έτσι και η κοινή γνώμη και οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι στη λήψη αποφάσεων θα αντιληφθούν ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί αυτό το 0,7 του ΑΕΠ μέχρι το 2015. Ε, αυτό δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το πετύχουμε, αλλά είναι άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε αργότερα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, περίμενα να λάβουν το λόγο πρώτα οι φιλελεύθεροι. Να ευχαριστήσω τον κύριο και για την εξαιρετική του προσπάθεια να καταγράψει και να εκθέσει το πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει αποσαφινιστεί αρκετά. Ρώτησα τον κύριο Πίμπαλξ τι σημαίνει μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς. Σκοπίμως έκανα την ερώτηση. Εγώ διάβασα την αιτιολογική σας έκθεση, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί. Αν αυτό είναι το νέο όρομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, στα πλαίσια των αναπτυξιακών πολιτικών και ορισμό σημαίνει ε, ναι ανάπτυξη, αλλά όχι ανάπτυξη που θα μετριέται σε ποσά ή ποσοστά, αλλά μιλάμε και για άλλα πράγματα. Πώς θα τα μετρήσουμε σε 10-15 χρόνια. Πώς θα μετρήσουμε την επιτυχία. Δεν νομίζω ότι είναι έξυπνα διατυπωμένη προσέγγιση και επίσης αποτελεί πρόβλημα συνολικότερης προσέγγισης επίσης. Δεν αναφέρομαι στην εκθεσή σας κύριε Κάσμαρκα, αλλά στο γεγονός ότι ο κύριος Πίμπαλξ μιλάει τώρα για νέο όραμα. Γιατί εμείς τώρα είμαστε μέσα στην οικονομική κρίση. Όλες οι χώρες διστάζουν να είναι πολύ γενναιόδορες στα αναπτυξιακά κονδύλια. Οπότε όταν μιλάμε για ε, αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων, ίσως ε, αυτό να έχει να κάνει και με την ασάφεια, δηλαδή μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς. Δεν θα πρέπει αυτό. Θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο, να μην ε, είναι αυτό ένα πρότυπο για το μέλλον. Από τη δική μου την πλευρά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάτς για την προσπάθεια που έκανε να μας υποβάλει ένα σχέδιο έκθεσης. Πάνω στη βάση αυτή όλοι και οι σκιώδεις και οι υπεύθυνοι των ομάδων μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε περαιτέρω διευκρινήσεις. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο αυτό που μας, σε αυτά, δεν είναι τόσο αυτό που μας είπε ο κύριος Κατσμάρκ, αλλά σε σχέση με την πράσινη βίβλο και το έγγραφο συζήτησης της Κομισιόν. Το πρόβλημα έχει να κάνει με την μελλοντική ανακοίνωση της Κομισιόν, γιατί δημιουργούνται μεγάλες ανασφάλειες. Ανακοίνωση η Κομισιόν ότι με το έγγραφό της Κατά πάσα πιθανότητα το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί στην κοινή γνώμη, ανεβλήθη η δημοσίευση του εγγράφου και νομίζω ότι αν δούμε τις δύο μελέτες που λάβαμε σήμερα για μια νέα ενωσιακή αναπτυξιακή πολιτική με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αν συγκρίνουμε τα δύο αντίτυπα, γερμανικά και αγγλικά βλέπουμε ότι αναδεικνύεται το πρόβλημα γιατί το ζητούμενο είναι αυτή η οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμού που μεταφράζεται γερμανικά ως ευρύτερη μεγέθυνση και στο εξώφυλλο αναφέρεται η ευρύτερη οικονομική μεγέθυνση ε, μεγαλύτερη μεγέθυνση μιλάμε για μια οικονομική μεγέθυνση που δεν έχει αποσαφινιστεί από τη συζήτηση. Τι ακριβώς πρέπει να γίνει με τη μεγέθυνση. Θα συμπεριληφθούν όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια μορφή ανακατανομή από τα πάνω προς τα κάτω ή θα είναι μια πρόσθετη οικονομική μεγέθυνση που θα φροντίσει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την καλύτερη κοινωνική πολιτική. Υπάρχουν λοιπόν από την αρχή κάποιες ασάφειες. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω και νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα η Κομισιόν γιατί οι υπεκφυγές δεν μας βοηθάνε το δεύτερο θέμα που θέλω να δείξω είναι το εξής. Σε διάφορες ε, ε, διατυπώσεις του κυρίου Κατσμάρεκ διαβλέπω τη δυνατότητα να καταθέσουμε τροπολογίες για να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Ίσως και μέσα από συζητήσεις με τον κύριο Κατσμάρεκ να δούμε αν η προσέγγιση η δική του συμβιβάζεται με τη δική μου και με τον άλλον. Καλό είναι λοιπόν να συντονιστούμε λίγο. Αναφέρομαι και στην καταπολέμη το κομμάτι που αναφέρεται στη φτώχεια και εδώ θα πρέπει να συνεννοηθούμε προς τα που θα κινηθούμε και από τη δική μου την πλευρά θα καταθέσω τροπολογίες οπωσδήποτε που σκοπό έχουν να προωθήσουν ε, τις δημόσιες υπηρεσίες, ε, δημόσιες κρατικές δομές, γιατί πέρα από την ιδιωτική οικονομία αυτό είναι πολύ σημαντικό στην αναπτυξιακή πολιτική και δεν μπορούμε να το βάζουμε στο περιθώριο. Επίσης, σε αυτά τα πλαίσια θα θέσω πάλι το ζήτημα της υποστήριξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών με βάση τη συνένεση της Ουάσιγκτον γιατί νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για να διορθώσει την στρεβλή ανάπτυξη των περασμένων ετών. Ο Γκερέντς και μετά η Κομισιόν. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω ε, μια γνώμη ως προς την έκθεση Κασμάρεκ και να μιλήσω για το θέμα της ανάπτυξης χωρίς περιορισμούς, χωρίς αποκλεισμούς. Έχετε δίκιο όταν μιλάτε για το θέμα της ερμηνείας αυτού του όρου. Δηλαδή, ε, τι εννοούμε, ότι στη μία περίπτωση γίνονται αποκλεισμοί, στην άλλη δεν γίνεται. Δεν Πώς το εννοούμε αυτό το inclusive. Όταν μιλάω για αποκλειστική ή επιμεριστική ή που αποκλείει μερικούς, σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει τους φτωχούς. Δεν προορίζεται σε αυτούς. Ενώ όταν μιλάμε για inclusive, μιλάμε για, χωρίς, για μία ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και η παγκοσμιοποίηση παράγει φτωχούς παντού και στις υποανάπτυξη χώρες και παντού γενικότερα. Και αυτό είναι το ουσιώδες ζήτημα στη συνεργασία, στην αναπτυξιακή συνεργασία. Ποια ομάδα φτωχών θα αντιμετωπίσουμε με αυτή την οικονομική αναπτυξιακή συνεργασία. Αυτό αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. Θα καταπολεμήσουμε τη φτώχεια σε χώρες που ήδη καταβάλουν, που, δεν έχουν τα μέσα να την καταπολεμήσουν ή σε χώρες που θα μπορούσαν να το κάνουν. Θα πρέπει το, πρώτα να επικεντρωθούμε στις φτωχές χώρες, τις λιγότερο αναπτυγμένες και μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και άλλα μέσα για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θα πρέπει να το κάνουμε και στη δική μας, στις δικές μας χώρες. Μιλάμε για φορολογική πολιτική, κοινωνική πολιτική υγείας. Μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής αλληλεγγύης. Όταν μιλάμε για βελτίωση και αποτελεσματικότητα, εδώ δεν μπορώ παρά να πω ότι προσυπογράφω. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον πολύπλοκο χαρακτήρα της φτώχειας που είναι απότοκη της παγκοσμιοποίησης και βλέπουμε ότι η κατανομή ακόμα και της φτώχειας είναι ιδιαίτερα άδικη. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Θα ήθελα να είναι ιδιαίτερα σύντομη θα πρέπει να τηρήσουμε το, το χρόνο, την προθεσμία μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, και εμείς συγχαίρουμε τον κύριο Κατσμάρκ για την έκθεση του Κομισιόν. Υποστηρίζει πολλά από αυτά που μας ανέφερε. Διαδικαστικά έχει τεθεί ένα θέμα χρονοδιαγράμματος. Πράγματι η ανακοίνωση μετά την πράσινη βίβλο προβλέπεται για το 3ο τέταρτο του 11, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, ίσως και αρχές Σεπτεμβρίου. Ως προς την ουσία τώρα, τα θέματα που αφορούν την συμπεριληπτική λεγόμενη ανάπτυξη προβλέπεται η ανακοίνωση να εξηγεί πιο σαφώς τι ακριβώς εννοεί ο όρος αυτός και είπε και ο Επίτροπος προηγουμένως μερικά. Καταρχήν, δηλαδή, θα πρόκειται για μια ανάπτυξη όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να ωφεληθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι φτωχοί και δεύτερον, θα υπάρχει σωστή κατανομή των αποτελεσμάτων της. Αυτά είναι τα κυριότερα στοιχεία. Το ένα πιο διαδικαστικό, δηλαδή οι διάφορες κοινωνικές ομάδες και οι διάεση φτωχοί θα μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και δεύτερον ως το, προς το αποτέλεσμά της θα κατανέμεται πιο δίκαια η ανακοίνωση λοιπόν αυτή θα προσπαθήσει να αναφέρει έναν πιο λεπτομερή ορισμό της έννοιας που δεν είναι όμως ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης γενικότερα. Ο στόχος είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Θα δούμε εμείς πώς μέσω μιας αναπτυξιακής πολιτικής ιδιαίτερα δε δημοσιονομικής βοήθειας επειδή η αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη βοήθεια γιατί πρόκειται και για άλλους τομείς πρέπει να δούμε πώς η αναπτυξιακή πολιτική και η βοήθεια μπορούν να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες για να δημιουργήσουν περισσότερη ανάπτυξη και εξάλληψη της φτώχειας. Ευχαριστούμε πολύ για τις αποσαφηνήσεις αυτές. Σας υποθυμίζω ότι η διορία κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 14 Απριλίου στις 6 ε, ώρα το απόγευμα ακριβώς. Ben, je sais pas. Il paraît que les Verts demander. Οι πράσινοι λέει ήθελαν παράταση, άμα δεν το ζητήσουν δεν θα δοθεί, δεν το ζητούν. Περνάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο Μήπως Παρασκευή το μεσημέρι στις 12 είναι δυνατόν. Παρασκευή στις 12 έχουμε έτσι λίγο περισσότερο χρόνο. Όχι αύριο, αλλά Παρασκευή στις 12. Καλά! Ορίστε. Άτε. Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην ε, αποστολή επιτήρησης των εκλογών στην Ουγγάντα. Ο κύριος Εδουάρδος Σικλούνα θα μας μιλήσει. Ήταν αρχιπαρατηρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι ο κύριος Σικλούνα, α, νάτος, νάτος. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Στις 5.30 έχουμε ψηφοφορία στην Επιτροπή, πολύ σημαντικές και πρέπει να φύγω. Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στις 18. Ήταν επιτυχής η αποστολή με ομαδικό πνεύμα με 120 συμμετέχοντες και πολύ, καλή, πολύ καλές σχέσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας συνήντησαν λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και παρέμειναν και μια-δύο μέρες μετά. Ευχαριστώ τον κύριο Ζέλερ προσωπικά που συνεργάστηκε και στην έκθεση και που μου επέτρεψε να έρθω έγινε μια αλλαγή κατά μία μέρα για να προλάβω κι εγώ το πρόγραμμά μου. Η αποστολή οργανώθηκε κάπως αργά, μια εβδομάδα πριν όμως όλοι ήταν στη θέση τους και διοργανώθηκε συνέντευξη τύπου. Όπως συνηθίζεται στη συνέντευξη τύπου μια εβδομάδα πριν υπάρχουν πιέσεις από τα μέσα ενημέρωσης για να μάθουν από εμά αν θέλουμε να κάνουμε σχόλια σχετικά με τα τεκτενόμενα εκεί. Και συνήθως δεν το κάνουμε αυτό, γιατί εμείς δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στην ίδια την εκλογική διαδικασία, αλλά παρακολουθούμε μόνο. Η πιο σημαντική πρώτη έκθεση ε, έγινε για τις εκλογές μία μέρα μετά και πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που έγινε την Κυριακή και οι πρώτες παρατηρήσεις μας ως εξής. Ε, η, πλήρη, ε, ε, η πλήρης έκθεση θα υποβληθεί αργότερα τη βδομάδα 2 με 5 Μαΐου μετά το Πάσχα. Σύνοψη συμπερασμάτων. Καταρχήν το benchmark που θα χρησιμοποιηθεί ποιο θα είναι για να αξιολογήσουμε τα στάνταρ των, των εκλογών. Είναι πολύ δύσκολο να το κρίνουμε αυτό γιατί ο ντόπιο πληθυσμός δεν απαντά σε σχόλια ναι ή όχι, ε, αν ήταν ελεύθερες και δίκαιες ή όχι. Και δεν είναι η πρόθεσή μας να επεκταθούμε. Εμεί θέλουμε να παρακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες, ε, τα, ε, τη, στάση των θεσμικών οργάνων κλπ. Πιστεύουμε ότι σε σχέση με τις εκλογές του 2006 υπήρξαν βελτιώσεις γιατί δεν υπήρχε γενικευμένη βία αν και υπήρξαν κάποια ε, επεισόδια. Το βασικό μας όμως πρόβλημα είναι όχι, το, το βασικό θέμα ήταν ότι υπήρξε βελτίωση και το είπαμε. Το απογοητευτικό είναι αυτό που αναφέρομαι ως ε, είναι οι διοικητικές αποτυχίες, η ε, ε, διοικητική μέρημνα δηλαδή που δεν επέτρεψε καλύτερη συμμετοχή στις εκλογές. Το δεύτερο ήταν είναι ότι το ένα δεύτερο θέμα είναι ότι δεν εξασφαλίστηκαν ε, ίσοι όροι παιχνιδιού μεταξύ υποψηφίων και πολιτικών κομμάτων. Καμιά φορά δεν διαφοροποιούνται τα δύο και πολλές φορές ε, έγιναν υπερβολικές δαπάνες ε, και αυτό το είδαν και οι παρατηρητές που ήταν εκεί για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα επεισόδια βίας ήταν σποραδικά, γενικά πιστεύουμε πάντως ότι ήταν ε, ειρηνικές εκλογές, ε, ήταν ε, περιορισμένοι οι λόγοι, οι επιδόσεις της αστυνομίας της Ουγγάντας έχει βελτιωθεί και αυτό το παρατηρήσαμε τη στάση τους. Υπήρχε έλλειψη εμπιστοσύνη στην εκλογική επιτροπή που είναι η ίδια επιτροπή εκλογών που είχε συσταθεί στις προηγούμενες εκλογές. Υπήρχε μεγάλη λογοκρισία από όλους τους εμπλεκομένους και δεν υπήρχε καθόλου εμπιστοσύνη προς αυτήν. Αυτό δημιουργήσε πολλά προβλήματα. Κάναμε πολλές συζητήσεις μαζί τους και τους τονίσαμε κάποια πράγματα που θεωρούσαμε ότι σίγουρα θα δημιουργούσαν προβλήματα και αυτό έγινε. Γι' αυτό είπαμε ότι ήταν δυνατόν να αποφευχθούν αυτά τα θέματα. Ε, τα εκλογικά μητρώα ε, δεν ήταν πλήρη και δεν υπήρχαν ταυτότητες που θα ήταν υποχρεωτικό να επιδεικνύουν οι ψηφοφόροι. Και αυτό οδήγησε σε προβλήματα. Κάποια ονόματα δεν υπήρχαν ή στέλναν μερικούς σε άλλα εκλογικά τμήματα ε, και δεν ήταν, εκεί, ούτε, δεν ήταν ούτε εκεί τα ονόματά τους πολλά προβλήματα αναγνώρισης ταυτοποίησης των ανθρώπων με βάση θολές φωτογραφίες. Άλλα προβλήματα αφορούν το εξής. Σχεδόν καμιά από τις βασικές συστάσεις του προκατόχου μου το από το 2006 δεν λήφθησαν υπόψη από την Επιτροπή των Εκλογών και αυτό ήταν απογοητευτικό. Τώρα τα καλά νέα είναι τα τα δικαστήρια τα οποία ε, είχαν πολλή δουλειά και ανταποκρίθηκαν καλά και επίσης το θέμα των... Ε, της εκπαίδευσης ε, ε, αυτό παλιά υπήρχε, ε, δημιουργούσε προβλήματα στην οργάνωση των εκλογών, το στήσιμο της κάλπης κλπ. Αυτά βελτιώθηκαν. Επίσης η εκπροσώπηση των, της αντιπολίτευσης ήταν προβληματική και δεν τα τόνιζε τα προβλήματα. Επίσης ήταν απογοητευτικό ότι είδαμε μεγάλη ανισορροπία στην ε, προσώπευση και την προβολή στα αποταμιμίε του ε, κόμματος της κυβέρνησης, του κυβερνητικού κόμματος και της αντιπολίτευσης. Η Ουγγάντα μπορεί να τα καταφέρει με βάση τις συστάσεις που διατυπώσαμε και στην έκθεσή μας και περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν όλα αυτά, θα εφαρμοστούν τις συστάσεις μας. Ευχαριστώ. Έχουμε καθυστερήσει γιατί πρέπει να συνεδριάσουν οι συντονιστές. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Νίλσεν, μετά στην Επιτροπή και όλα αυτά θα γίνουν σε 7 λεπτά. Ευχαριστώ εντάχει. Είμαι εδώ γιατί ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας ε, για ε, τις εκλογές στην Ουγγάντα. Ο κύριος Σικλούνα επέμεινε σε ένα σημείο που για μένα είναι σημαντικό και λυπηρό. Δηλαδή οι συστάσεις που έγιναν το 2006 δεν ελήφθησαν υπόψη, δεν ε, θα ήθελα να επεκταθώ, είναι πολύ ανησυχητικό το θέμα και θα ήθελα να πω ότι με εξέπληξε το ανακοινοθέν της ΥΠΑ της εκπροσώπου στις 20 Φεβρουαρίου για τις εκλογές στην Ουγκάντα. Απευθύνθηκα στην ΕΙΕΒ και θα μου δοθεί αύριο απάντηση στην ε, Νομική Επιτροπή, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αυτή η προεκλογική διαδικασία ε, είχε, ε, γνώρισε πολύ αρνητικά συμβάντα όπως εκφοβισμούς και ούτω καθεξής και λυπάμαι γιατί είπα ότι εκπρόσωπος δεν έλαβε υπόψη τη γνωμοδότηση της αντιπροσωπείας, δηλαδή δεν έλαβε υπόψη τη γνώμη της αποστολής παρατήρησης της εκλογικής ε, διαδικασίας γιατί χρειάστηκε να μεταβούμε για αρκετές εβδομάδες σε αυτή τη χώρα και νομίζω ότι στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν οι υπόψη οι διαπιστώσεις μας. Εγώ ήρθα εδώ για να σας το πω γιατί με ξέπληξε το γεγονός ιδιαίτερα τη στιγμή που αμφισβητούμε αυταρχικά καθεστώτα ανά, αυτό, ανά τον κόσμο. Λυπάμαι για τη συγκάλυψη αυτού του αυταρχικού καθεστώτος από την ύπατη εκπρόσωπο. Ναι, θα έπρεπε να είναι εδώ κάποιος εκπρόσωπος η ε.ε.δ. αλλά δεν είναι. Και άρα το λόγο έχει επιτροπή. Ποιος θα λάβει το λόγο. Ως προς το τελευταίο. Γι' αυτό το τελευταίο που είπατε, νομίζω ότι θα σας δοθεί λεπτομερέστερη απάντηση γιατί κάνατε την ερώτηση. Αλλά δύο πράγματα πρέπει να πούμε. Πρώτον, υπάρχει διαφορά μεταξύ της δήλωσης της κυρίας Άστον, που είναι γενική δήλωση, και υπάρχει και η δήλωση των παρατηρητών που είναι σχετικά λεπτομερής δήλωση. Είναι λοιπόν μια διαφορά αυτή που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Δεύτερον, επί της ουσίας αυτό τώρα περισσότερο. Εμείς είμαστε ευτυχείς διότι μειώθηκε πολύ η βία. Υπήρχε πολύ λιγότερη βία αυτή τη φορά από ό,τι την προηγούμενη. Στις προηγούμενες, ε, τις τελευταίες εκλογές ε, είχε ε, συλληφθεί ο επικεφαλής αντιπολίτευσης τρεις μήνες πριν. Και αυτό βέβαια επηρέασε πολύ την ισότητα των υποψηφίων. Επίσης ήταν η δεύτερη πολυκομματική διοργάνωση εκλογών στην Ουγγάντα. λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και την ε, βλέποντας με ιστορική προοπτική το θέμα, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος. Κύριε Ντέπα, εντάχει Ήξερα τον πρόεδρο για 20 περίπου χρόνια και είχε συσταθεί και ένα Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης. Για πολλά χρόνια έγινε προσπάθεια ε, εκλογών με συμμετοχή πολλών κομμάτων, αλλά δεν ε, πίστευε ότι θα μπορούσε να ακολουθηθεί το πρότυπο του Westminster στην Αφρική. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση στη Βρετανία κατά πώς θα πρέπει να επιβάλλουμε αυτή τη δυτική ιδέα στην Αφρική ή κατά πώς θα πρέπει να αφήσουμε την Αφρική να ακολουθήσει το δικό της πρότυπο. Ο πρόεδρος για 20 χρόνια προσπάθησε να το επιβάλλει αυτό. Εάν λοιπόν δέχονται αυτό το δυτικό πρότυπο πολιτικής, ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εδώ επισέρχεται και ένα στοιχείο εκπαίδευσης και θα πρέπει να γίνει πολύ ε, μεγάλη εργασία. Εγώ προσπάθησα να πείσω τον Πρόεδρο ότι έτσι θα πρέπει να προχωρήσει και είπε ότι υπάρχουν επτά διαφορετικά συμβούλια και δεν υπάρχει αντιπαράθεση στην Ουγγάντα. δεν υπάρχουν πρότυπα αντιπαράθεσης. Βεβαίως είναι στην εξουσία πολλά χρόνια, υπερβολικά πολλά χρόνια αλλά θα πρέπει να διδάξουμε του, τον πληθυσμό της Ουγκάντα ότι ε, ε, εμείς έχουμε διαφορετικό πρότυπο και δεν έχουν άλλη επιλογή. Με τα αποτελέσματα που πολύ καλά γνωρίζουμε του δικού μας του μοντέλου. Λοιπόν, στις 2 Μαΐου θα γίνει η προσεχής ε, συνεδρίασή μας από τις 3 στις 6.30. Θα συνεχίσουμε εδώ με τους συντονιστές. Κύριε Ντέβα, ελάτε εδώ γιατί εγώ πρέπει να φύγω. Και θα ήθελα οι συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα, οι άλλοι να αποχωρήσουν και να συζητήσουν, να συνεχίσουν τα πηγαδάκια τους. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε αυτή τη συνεδρία και θα τα πούμε σύντομα. Χαίρετε.